Καλησπέρα. Υπάρχουν κάποια προβλήματα με τις μεταφορές σήμερα. Οπότε φαντάζομαι θα έρθουν και οι υπόλοιποι σιγά σιγά. Έχουμε το σχέδιο μερίσιας διάταξης. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ. Έγκριση των πρακτικών. Πρόκειται για τη συνεδρίαση της 28 η Νοεμβρίου του 2013 έχουν διανεμηθεί και δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα καμιά αντίρρηση. Συνεπώς, θεωρώ ότι εγκρίνονται. Τις ανακοινώσεις της Προέδρου ως ήθιστε θα σας ε, τις κάνω στην ψηφοφορία. Και έτσι φτάνουμε στο σημείο 4, που είναι ο διάλογος επινομισματικών θεμάτων με τον Μάριο Ντράγκη, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ως ήθιστε, θα έχουμε πρώτα μια παρουσίαση από τον ίδιο τον κύριο Ντράγκη και στη συνέχεια 5 λεπτά ερωτήσεις και απαντήσεις. Αν ε, πέντε λεπτά ξοδέψετε, δεν έχετε απάντηση. Αν ε, ένα λεπτό, τότε θα έχετε απάντηση για τέσσερα λεπτά. Λίγο πολύ έτσι πάει. Συνεπώς, χαίρομαι που είσαστε εδώ, Μάριο. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, σε ευχαριστώ Σάρον, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Είναι πραγματική χαρά για μένα να βρίσκομαι στην Επιτροπή σας σε μια τόσο αποφασιστική στιγμή. Τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες, μέχρι το τέλος της νομοθετικής αυτής θητείας, θα είμαστε σε θέση να δείξουμε αν η Ευρωζώνη τελικά μπορεί να κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προ την Τραπεζική Ένωση. Εγώ πιστεύω ότι το δικό σου θεσμικό όργανο μπορεί να διαδραματίσει έναν σημαντικό και επικοδομητικό ρόλο, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι το επόμενο αυτό βήμα θα οδηγήσει και θα έχει ουσιαστικά μια πραγματικά ευρωπαϊκή διάσταση. Είναι η τελευταία επίση φορά που θα συζητήσω μαζί σα με κάθε δυνατή λεπτομέρεια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον νέο εποπτικό μηχανισμό. Περιμένουμε να διορίσει το Συμβούλιο επίσημα την κυρία Ντανιέλ Νουή, η οποία θα γίνει η επικεφαλής του Εποπτικού Συμβουλίου από την 1η Ιανουαρίου του 2014. Και στη συνέχεια θα γίνει η βασική συνομιλητριά σας σε σχέση με τον ε, ενιαίο ε, μηχανισμό εξυγίανσης. Σήμερα θα εξετάσουμε καταρχάς τις οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη και στη συνέχεια θα μπορέσω να σας παρουσιάσω ακόμα περισσότερο κάποιες αποφάσεις που έχουμε πάρει στα πλαίσια της νομισματικής μας πολιτικής και θα σας παρουσιάσουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί προκειμένου να θεσπίσουμε τον ε, ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης. Από την ε, συνεδρίαση που είχαμε το Σεπτέμβριο και στο ενδιάμεσο διάστημα οι πληροφορίες οι οποίες μας έφτασαν πραγματικά επιβεβαίωσαν ότι οι πιέσεις στις τιμές παραμένουν υποτονικές στο μεσοπρόθεσμο διάστημα. Η οικονομική ανάκαμψη στην Ευρωζώνη είναι ιδιαίτερα έφραστη. Το πραγματικό ΕΠ στην Ευρωζώνη επεκτάθηκε τα τελευταία δύο τρίμηνα από τον Ιούλιο στο Σεπτέμβριο, αυξήθηκε κατά 0,1% από το ένα τρίμηνο στο άλλο και σε συνέχεια κατά 0,3% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2013. Οι εξελίξει όσον αφορά του δείκτε εμπιστοσύνη μέχρι τον Νοέμβριο καταδεικνύουν ότι έχουμε μία μικρή ανάπτυξη και αύξηση το τελευταίο τρίμηνο του έτου. Παράλληλα, τα ποσοστά ανεργία παραμένουν υψηλά. και πρέπει να γίνουν οι απαραίτητε προσαρμογέ στου ισολογισμού του χρηματοπιστωτικού και μη χρηματοπιστωτικού τομέα. Και οι ισολογισμοί αυτοί πειράζουν πάρα πολύ την οικονομική δραστηριότητα. Εξετάζοντας το απότερο μέλλον, περιμένουμε ότι η παραγωγή θα συνεχίσει να ανακάμπτει με αργό ρυθμό. Αυτό οφείλεται κυρίω σε κάποιε βελτιώσει που έχουν γίνει όσον αφορά την εγχώρια ζήτηση, η οποία υποστηρίζεται από τη δική μα προσαρμοστική νομισματική πολιτική, σε σχέση με τη ζήτηση δηλαδή. Θα πρέπει επίση η Ευρωζώνη στο μέλλον να ωφεληθεί όλο και περισσότερο από μια ενδυνάμωση τη ζήτηση για εξαγωγέ η βελτίωση επίση των συνθήκων στι χρηματοπιστωτικέ αγορέ, καθώ επίση και η μείωση τη αβεβαιότητα, από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά περνάει και στην πραγματική οικονομία. Τέλο, η πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη δημοσιονομική εξυγίανση έχει ενισχύσει την εμπιστοσύνη των αγορών όσον αφορά την ανθεκτικότητα τη Ευρωζώνης. Και αυτό με τη σειρά του θα πρέπει να επηρεάσει θετικά την ανάκαμψη. Ωστόσο, οι κίνδυνοι όσον αφορά τις μελλοντικέ μα προοπτικές υφίστανται και έχουν να κάνουν κυρίως με κάποιες εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία καθώς επίσης και στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές. Υψηλότερες ε, τιμές για κάποια προϊόντα, χαμηλότερη ζήτηση για κάποιες εξαγωγές, καθώς επίσης και μη επαρκείς διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε κάποιες χώρες Ευρωζώνης θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις οικονομικές προϋποθέσεις, οικονομικές συνθήκες ο ετήσιο πληθωρισμό συναρρισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή αυξήθηκε τον Νοέμβριο κατά 0,9% σύμφωνα με τι εκτιμήσει τη ε, Eurostat, μετά από μια πολύ έντονη πτώση τον Οκτώβριο σε 0,7%. Οι ε, συνεχιζόμενες πιέσεις στις τιμές στην Ευρωζώνη θα παραμείνουν υποτονικές ε, κατά το μεσοπρόθεσμο διάστημα ενδεχομένως να βιώσουμε μια παρατεταμένη περίοδο χαμηλού πληθωρισμού, η οποία θα ακολουθηθεί στη συνέχεια από μια αυξητική τάση προς πληθωρισμό που θα βρίσκεται κάτω ή κοντά στο 2% αλλά σε ένα μεταγενέστερο διάστημα αυτό. Αυτό δικατοπτρίζει την αργή, τον αργό ρυθμό της ανάκαμψης καθώς επίσης και το ότι ο μεσοπρόθεσμος πληθωρισμός παραμένει συναρτισμένος με την εξέλιξη των τιμών, καθώς επίσης και με τη δική μας πολιτική σταθερότητα των τιμών. Η δυναμική επίσης των πιστώσεων παραμένει υποτονική. Ο ετήσιος ρυθμός δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα έχει σταθεροποιηθεί σε αρνητικά επίπεδα. Επίσης έχουμε χαμηλή δυναμικότητα όσον αφορά τα δάνεια, τα οποία αντικατοπτρίζουν τον υφιστάμενο, τις υφιστάμενες συνθήκες που ισχύουν στους επιχειρηματικούς κύκλους, καθώς επίσης και τους υψηλούς κινδύνους που ακόμα σχετίζονται με την δανειοδότηση, με τις πιστώσεις. Θα ήθελα τώρα να σας παρουσιάσουμε περισσότερες λεπτομέρειες τις πιο πρόσφατες αποφάσεις που έχουμε λάβει στον τομέα της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής. Τον Ιούλιο του 2013 αρχίσαμε να εφαρμόζουμε το πρόγραμμα λεγόμενο Forward Guidance, που έχει να κάνει με τις μελλοντικέ προοπτικές της νομισματικής μας πολιτικής, εν ιδιαίτερα σταθές περιβάλλον. Είχαμε πει τότε ότι περιμέναμε ότι τα βασικά επιτόκια θα παραμένανε στα τωρινά ή ακόμα και σε χαμηλότερα επίπεδα για ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η δήλωση αυτή εξαρτιόταν από μια γενικότερη υποτονική εξέλιξη του πληθωρισμού και για το μεσοπρόθεσμο διάστημα, πράγμα το οποίο επιβεβαιώθηκε όπως εξήγησα πριν από λίγο. Σύμφωνα λοιπόν με τις προβλέψεις μας αυτές αποφασίσαμε τον Νοέμβριο να μειώσουμε τους ε, βασικούς ε, δείκτες, τα βασικά επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ακόμα περισσότερο. Τα βασικά επιτόκια για τις ε, δράσεις αναχρηματοδότησης μειώθηκαν κατά 25 μονάδες σε 0,25% και οι δείκτες όσον αφορά το περιθώριο δανεισμού μειώθηκαν στο 0,7%. Δεν αλλάξαμε καθόλου όμως το ποσοστό όσον αφορά τις, ε, τα επιτόκια καταθέσεων. Συνεχίζουμε βέβαια τις ε, προπτικές μας. Συνεχίζουμε να ακολουθούμε αυτές τις νομισματικές προπτικές και θεωρούμε ότι τα βασικά επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα παραμείνουν σε ένα χαμηλό επίπεδο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατά αυτόν τον τρόπο η νομισματική μας πολιτική θα εξακολουθήσει να είναι προσαρμοστική για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί. Η προσαρμογή των επιτοκίων όμω από μόνη τη δεν αρκεί προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα των τιμών. Και όταν αναφέρομαι σταθερότητα των τιμών, ουσιαστικά αναφέρομαι σε σταθερότητα προ τι δύο κατευθύνσει. Κατά τη διάρκεια της ε, κρίσης αυτής είδαμε ότι η μείωση των επιτοκίων έχει ε, περάσει όλο και πιο αργά και ανώμια ουσιαστικά στις διάφορες χώρες της Ευρωζώνης εξαιτίας του κατακαιρματισμού των χρηματοπιστωτικών αγορών. Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό, εγκρίναμε τελευταία χρόνια μια σειρά από μη συμβατικά μέτρα. Στόχος μας ήταν και παραμένει να έχουμε μια πιο αποτελεσματική μετάδοση, διάχυση των επιτοκίων τη μείωση των επιτοχίων τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου η νομισματική μα αυτή πολιτική να καταφέρει πραγματικά να φτάσει στι εταιρείε και τα νοικοκυριά τη Ευρωζώνη. Και για αυτόν τον λόγο αποφασίσαμε το Νοέμβριο να συνεχίσουμε να κάνουμε όλες τις δραστηριότητες αναχρηματοδότησης με τον ίδιο ακριβώ τρόπο και με τα ίδια επιτόκια τα οποία εφαρμόζουμε αυτή τη στιγμή μέχρι τον Ιούλιο του 2015. Κατά αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να ελαφρώσουμε κάπω τα προβλήματα χρηματοδότηση ε, των τραπεζών τα οποία διστάζουν αυτή τη στιγμή να δανείσουν προ εταιρείε και νοικοκυριά. Πριν από δύο χρόνια καταφέραμε να στηρίξουμε τη χρηματοδότηση των τραπεζών μέσω μακροπρόθεσμων ε, δραστηριοτήτων χρηματοδότησης σε μια τριετή χρονική περίοδο. Καθότι βελτιώθηκε η κατάσταση χρηματοδότησης τραπεζών έκτοτε, οι τράπεζες φέτος είναι σε θέση να αποπληρώσουν περίπου το 40% του αρχικού ποσού που τους είχε δοθεί. Έτσι λοιπόν, η υπερβολική ρευστότητα στις χρηματαγορές αρχίζει σιγά σιγά και μειώνεται. Παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς τις επιπτώσεις που εξελίξει αυτές θα μπορούσαν να έχουν στην νομισματική μας πολιτική. Και είμαστε βέβαια πάντα έτοιμοι να εξετάσουμε και άλλα εναλλακτικά διαθέσιμα μέσα. Ο συνήθως απαιτείται κάποιος χρόνος προτού δούμε τα πραγματικά αποτελέσματα της νομισματικής μας πολιτικής στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στην πραγματική οικονομία. Οι αποφάσεις που λάβαμε τον Νοέμβριο όσον αφορά τα επιτόκια, οι αποφάσεις όσον αφορά τις μελλοντικές μας προοπτικές, καθώς επίσης και τα επιτόκια τα οποία χρησιμοποιούμε για τις δραστηριότητες χρηματοδότηση, έχουν τελικά θετικές επιπτώσεις στην οικονομία. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν πραγματικά αναλάβει δεσμεύσεις υποπροϋποθέσεις προκειμένου να ακολουθήσουν τη δική μας προσαρμοστική νομισματική πολιτική. Τα επιτόκια όσον αφορά τις χρηματαγορές έχουν μειωθεί, καθώς επίσης και η απόδοση κάποιων τραπεζικών ομολόγων. Από την άλλη όμως γνωρίζουμε πλήρως ότι υπάρχει ένας κίνδυνος πτωτικής τάσης όσον αφορά το χαμηλό αυτό πληθωρισμό, μείωση αστικά της οικονομικής ανάπτυξης. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι έτοιμο, όπως το είπαμε άλλωστε και στην τελευταία συνέντευξη τύπου μας, να αναλάβει δράση να αυτό απαιτηθεί. Δεν βλέπουμε επίσης να υπάρχουν κίνδυνοι από χρηματοοικονομικές ανισορροπίες οι οποίες σχετίζονται με αυτό το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι υπάρχει μια γενικότερη υποτονική τάση όσον αφορά τις νομισματικές και πιστοτικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη. Ωστόσο, αν τελικά δημιουργηθούν τέτοιες ανισορροπίες, θα πρέπει να αναλάβουν δράση οι μακροπροληπτικές αρχές οι οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα μέσα αναγορά. Καταλαβαίνετε ότι οι τοπικοί κίνδυνοι πρέπει να αντιμετωπιστούν με τοπικά χρηματοοικονομικά μέσα. Γι' αυτόν τον λόγο οι εποπτικές αρχές όπως ε, ο ενιαίος μηχανισμός εξυγίανσης έχουν πλέον αυτά τα μέσα μικρό και μακροπροληπτικής ε, ε, πολιτικής και είμαι σίγουρο ότι θα χρησιμοποιηθούν τα μέσα αυτά εφόσον απαιτηθεί κάτι τέτοιο. Θα ήθελα τώρα να σα ενημερώσω για τι τελευταίε εξελίξει που είχαμε όσον αφορά τη δημιουργία του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού. Οι εσωτερικές μας προπαρασκευαστικές διεργασίες έχουν ως στόχο να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αναλάβει τις εποπτικές της αρμοδιότητε τον Νοέμβριο του 2014. Κατά αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσουμε ότι οι αρμοδιότητες νομισματικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως προς σταθερότητα των τιμών δεν πρόκειται να επηρεαστούν από κάποιες αποφάσεις που θα ληφθούν όσον αφορά την τραπεζική εποπτεία. Οι εσωτερικοί λοιπόν κανόνες αυτή τη στιγμή δημιουργούνται προκειμένου να διαχωρίσουμε την νομισματική πολιτική από, την εποπτική, από τις εποπτικές αρμοδιότητες. Οι μονάδε οι οποίε θα έχουν να κάνουν με την ε, λήψη αποφάσεων στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα είναι εντελώ ξεχωριστέ. Θα έχουμε μια τέτοια αρχιτεκτονική και οστερική δομή έτσι ώστε οι δύο αρμοδιότητε απλώ να ενημερώνονται, οι δύο μονάδε να ενημερώνουν μία την άλλη, χωρί να υπάρχει όμω καμία απολύτω σύγχυνση. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε επίση να έχουμε αλληλοεπικαλύψει στη δικασία λήψη αποφάσεων. Κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι αποδοτικό από οικονομική πλευρά και νομίζω ότι και εσεί θα είστε ικανοποιημένοι με κάτι τέτοιο. Όσον αφορά τώρα την πρόσληψη προσωπικού, έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία προκειμένου να προσληφθεί προσωπικό σε μέσο και ψηλό βαθμό επίπεδο. Περαιτέρω προσλήψεις θα γίνουν στο μέλλον. Στα πλαίσια των προετοιμασιών μας για τη νέα αυτή δομή, ασχολούμεθα ιδιαίτερα με την αξιολόγηση, προκειμένου να μπορούμε να έχουμε μια πραγματική αναθεώρηση και αξιολόγηση των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών, καθώς επίσης και μια καλύτερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε ένα υψηλότερο επίπεδο διαφάνειας και θα βελτιωθούν οι διαθέσιμες πληροφορίες. Επίσης, κατά αυτόν τον τρόπο θα διευκολυνθεί η ανάκαμψη του τραπεζικού τομέα και θα καταφέρουμε έτσι να εντοπίσουμε τις σωστές διορθωτικές δράσεις. Και επίσης, κατά αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί και απαραίτητη εμπιστοσύνη προς τις τράπεζες, εφόσον πλέον θα είναι υγιείς. Η όλη διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί λίγο προτού αναλάβει τις εποπτικές της δραστηριότητες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήδη διεξήγει κάποιες συνεδριάσεις τον Νοέμβριο στην Φραγκφούρτη με τις τράπεζες εκείνες οι οποίες θα περάσουν σε αυτό το καθεστώς της ε, συνολικής αξιολόγησης. Είχαμε πολύ θετική ανταπόκριση στις συζητήσεις αυτές και είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε μια πρώτη επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων προκειμένου να δούμε και ποιες είναι οι ερωτήσεις ή πληροφορίες που θέλουν να μας δώσουν οι τράπεζες αυτές. Επίσης εξηγήσαμε τότε ότι ε, είμαστε υπέρ του να αναλάβουν προληπτική δράση ήδη από τώρα οι τράπεζες προκειμένου να καταφέρουν να διορθώσουν τους ισολογισμούς τους, ιδίως όσον αφορά το μετοχικό κεφάλαιο. Επίσης, ε, περαιτέρω διεργασίες για την ε, συνολική αξιολόγηση λαμβάνουν χώρα προσπαθούμε να αρχίσουμε την όλη διαδικασία αξιολόγηση, ποιοτική αξιολόγηση των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών. Ήδη έχουμε αρχίσει να συλλέγουμε πληροφορίε προς προ αυτό. Επίση, προσπαθούμε να δούμε ποιε θα είναι ακριβώ οι παράμετροι οι οποίε θα χρησιμοποιηθούν για να γίνουν τα stress tests σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή στι αρχέ του 2014. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να σα εξηγήσω τι πρόκειται να γίνει με τα κρατικά ομόλογα. Στην Asset Quality Review προσπαθούμε να αξιολογήσουμε τα την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών και θα χρησιμοποιηθεί το εφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο. Δεν πρόκειται εμεί ω Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να τροποποιήσουμε το πλαίσιο αυτό το νομοθετικό. Γίνεται μια γενικότερη συζήτηση αυτή τη στιγμή και θεωρώ ότι ο κατάλληλο χώρο για οποιαδήποτε πρόταση είναι η Επιτροπή τη Βασιλεία. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι θα πρέπει στα πλαίσια των stress test να καλύψουμε πάρα πολλά στοιχεία του ενεργητικού τραπεζών και βέβαια ανάμεσα σε αυτά θα καλύψουμε και τα κρατικά ομόλογα. Προκειμένου να είναι αυστηρό όμω ο έλεγχο αυτό, θα πρέπει να υπάρχουν και τα απαραίτητα backstops, οι απαραίτητοι προστατευτικοί ε, μηχανισμοί, οι οποίοι θα πρέπει να αρχίζουν να ισχύουν και να λειτουργούν. Θα πρέπει να δούμε καταρχάς ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα μπορέσουν στα πλαίσια του bail-in να αναλάβουν δράση. Πρώτα θα πρέπει να απευθυνθούμε στους ιδιωτικούς πόρους και μόνο στο τέλος στον Ευρωπαίο ε, φορολογούμενο ή στις καταθέσεις. Τώρα, όσον αφορά την οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών. Είμαι σαφώς υπέρ της συμφωνίας που έχει επιτευχθεί και θεωρώ ότι θα αποτελέσει ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση Τραπεζικής Ένωσης. Ωστόσο, Προκειμένου η τραπεζική αυτή ένωση να είναι αξιόπιστη θα πρέπει να γίνει και κάτι ακόμα. Ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός χρειάζεται έναν ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης και θα πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητε αρμοδιότητε τόσο για την εποπτεία όσο και για την εξυγίανση και θα πρέπει δύο αυτέ αρμοδιότητε να ευθυγραμμιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεπώ, σα καλώ επιγόντω και εσά και το Συμβούλιο να δημιουργήσετε το ταχύτερο δυνατό έναν στεναρό ενιαίο μηχανισμό εξυγίανση σε καθάριση τραπεζών για τον οποίο απαιτούνται ουσιαστικά τα εξή ακόλουθα. Ένα ενιαίο σύστημα, μια ενιαία αρχή και ένα ενιαίο ταμείο. Δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο μηχανισμό εξυγίανσης, ε, ο οποίος να είναι μόνο κατόνομα ενιαίος, μόνο θεωρητικά ενιαίος. Ως προς λοιπόν αυτό, Φοβάμαι ότι η όλη διαδικασία λήψη αποφάσεων μπορεί να είναι πάρα πολύ πολύπλοκη και τελικά να μην επαρκούν οι απαραίτητε χρηματοπιστωτικέ διευθετήσει. Πάντω είμαι σίγουρο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη συνεργασία του Συμβουλίου θα δημιουργήσει μια πραγματικά αυθεντική τραπεζική ένωση. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα και προσβλέπω στι ερωτήσει σα. Ευχαριστώ πολύ συμφωνούμε για αυτά που λέτε όσον αφορά τον μηχανισμό εξυγίανσης όπως και μετά Τώρα, πρώτη ερώτηση από το ΕΛΚ. Ο Παύλος Ζέλβα. anyway. Είσαι ο πρώτος στον καταλόγο μου. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Δεν ήξερα ότι ήμουν ο πρώτος. Δύο πράγματα θέλω να ρωτήσω. Σε σχέση με δύο διαφορετικά ζητήματα, αλλά που έχουν σχέση μεταξύ τους. Για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πρώτα απ' όλα. Είσαστε ικανοποιημένος με τις επιπτώσεις που έχουν τα μέτρα που έχει οθετήσει μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Γιατί βλέπουμε ότι κάθε μήνα που περνάει σε ορισμένες χώρες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δυσκολεύονται ακόμα περισσότερο να έχουν πρόσβαση ε, σε χρήματα, σε δάνεια. Είναι μια συζήτηση που γίνεται λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τα μη συμβατικά μέτρα προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση αυτή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως ε, αντίστοιχα μέτρα υιοθέτησε η Τράπεζα της Αγγλίας. Έπειτα πάντα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά τον νέο μηχανισμό εξυγίανσης. Είπατε ότι πρέπει κανείς να είναι ισχυρός και αξιόπιστος. Από αυτά που είπατε εγώ αντιλαμβάνομαι πως η συμφωνία που ενέκρινε το Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα δεν είναι αρκετά ισχυρή και αξιόπιστη. Και αν είναι έτσι, πιστεύετε ότι υπάρχει περιθώριο λιγμών στο ΕΚΟΦΗΝ αυτή τη εβδομάδα προκειμένου να βελτιωθεί η συμφωνία αυτή. Τι προσδοκίες έχετε εσείς, Πρόεδρε, από αυτού. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δράγκη. Ευχαριστώ πολύ. Με ρωτάτε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι με τις διάφορες επιχειρήσεις LTRO που αρχίσαμε πριν από ένα χρόνο έχουμε ήδη αντιμετωπίσει σε ένα βαθμό τουλάχιστον τα ζητήματα αυτά και γενικότερα την οικονομία. Δεν έχουμε ξεχάσει ότι το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς είχαμε πάνω από 230 δισεκατομμύρια ομόλογα που οφείλονταν σε εκείνη την χρονική περίοδο. Και εμείς αυτό το αντιμετωπίσαμε. Στη συνέχεια διαπιστώσαμε μια πολύ αργή διαδικασία για να φτάσουν τα χρήματα αυτά στην πραγματική οικονομία. Οπότε η ερώτησή σας είναι γιατί δεν κάνουμε κι εμείς ό,τι κάνουν άλλες χώρες για την αναχρηματοδότηση. Κοιτάξτε, το πρόγραμμα αυτό έχει διάφορα, διάφορα στοιχεία. Το ένα είναι εγγύησει. και το θέμα της ρευστότητας. Είναι στοιχεία τα οποία ήταν παρόντα και στο αρχικό Long Term uh, Refinance Operation. Στο LTRO είπαμε στις τράπεζες ότι μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα δάνεια τα οποία έκαναν στους πελάτες τους ως εγγύηση για να μπορούν να δανειστούν στη συνέχεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άρα δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, τη χρηματοδότηση την συνδέσαμε με το θέμα των εγγύσεων. Τώρα το θέμα είναι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω. Ναι, το σκεφτόμαστε. Προβληματιζόμαστε πάνω σε αυτό, αλλά όλοι πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι περίπλοκη διαχείριση ενός τέτοιου συστήματος ε, σε 17-18 που να είναι χώρες. Είναι δύσκολο να λειτουργήσει. Δεν λειτουργεί με την ίδια ευκολία σε μια χώρα και σε 17 χώρες ένα τέτοιο πρόγραμμα. Πάντω τα χρήματα αυτά θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα φτάσουν στην πραγματική οικονομία και δεν θα σταματήσουν στι τράπεζε ή στα ομόλογα. Δεν υποτιμούμε βέβαια το γεγονός ότι πρόκειται για ένα περίπλοκο πρόγραμμα που συνεχίζουμε όμως να εξετάζουμε. Για το δεύτερο ζήτημα. Με ρωτάτε τι προσδοκίες έχω. Περισσότερο από προσδοκίες θα έλεγα ότι ο ε, μηχανισμός εξυγίανσης απαιτεί όλες οι πλευρές να λειτουργήσουν. Δηλαδή προκειμένου να έχουμε την Τραπεζική Ένωση και τη σωστή αντίληψη από πλευράς των αγορών, είναι απαραίτητο να υπάρχει μια καλή συμφωνία για τον νέο μηχανισμό εξυγένσης. Αυτό είναι κάτι αναγκαίο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η Ελίζα Φεραίρα εκ μέρους των Σοσιαλιστών τώρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε εδώ ανάμεσά μας για άλλη μια φορά. Θα μιλήσω αγγλικά για να εξαπλουστεύσω τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε ανάμεσά μας και είσαστε κοντά μας και σας ευχαριστώ για το έργο που επιτελέσατε να υπερασπιστείτε το ευρώ και την ευρωζώνη. Τρεις σύντομες ερωτήσεις έχω. Η πρώτη, η πρώτη αφορά το SRM. Είμαι η συγγήτρια και συμμερίζομαι το μήνυμά σας απόλυτα, αλλά θα ήθελα να διασφαλίσω από εσάς ή να μου πείτε εσείς αν μπορείτε να διασφαλίσετε ότι το SSM δεν θα καταλήξει να έχει μία δύο κατηγοριών αντιμετώπιση τραπεζών. Γιατί αν έχουμε δύο κατηγορίες αντιμετώπιση στο SSM, ανοίγουμε πύλες, πόρτες και παράθυρα όχι για ένα ενιαίο σύστημα, αλλά για ένα διαφοροποιημένο σύστημα. Δεύτερη ερώτηση, για το ESM γιατί όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση του SSM, υπήρχε η υπόσχεση ότι το ESM θα κατέληγε ανακεφαλαιώντας άμεσα, ανακεφαλοποιώντας άμεσα τις τράπεζες. Αυτό δεν συνέβη. Το σύστημα εξακολουθεί να βασίζεται σε εγγυήσεις από τα κράτη-μέλη που παρακολύει αυτό τον στόχο του να διαχωρίσουμε το κρατικό χρέος, δημόσιο χρέος από το τραπεζικό χρέος και να επιτευχθεί αυτή η διαφοροποίηση. Δεν έχει επιτευχθεί αυτή η διαφοροποίηση, αυτός ο διαχωρισμός και δεν έχει επιτευχθεί όταν προσπαθούμε να, να κινητοποιήσουμε την, την οικονομία μέσω των τραπεζών. Δεν υπάρχει λοιπόν αυτή η δυνατότητα. Αυτό απαιτεί λοιπόν μια νέα προσέγγιση στο θέμα πιθανότατα. Και αυτή είναι ακριβώς η ερώτησή μου επακριβώς. Ποιος είναι ο ρόλος λοιπόν του ESM ε και η τρίτη μου ερώτηση είναι οι επενδύσεις όσον αφορά την ζήτηση. Ένα από τα θέματα που δεν συμφωνώ είναι ε, σε σχέση με την Τρόικα. Η Τρόικα και οι εκπρόσωποι των τριμερών ήταν ε, ισχυρότατοι εκπρόσωποι αυτής της τάσης. Τώρα Κάποιες ε, χώρες ακολούθησαν τη συνταγή τυφλά στις τελευταίες φάσεις ε, του προγράμματος προσαρμογής. Τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Ποια μαθήματα μπορείτε να συναγάγετε από τη συμμετοχή σας στην τριμερή ή στις τριμερείς διαδικασίες. Το μεταβατικό πρόγραμμα. Με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα μπορέσει αυτό το μεταβατικό πρόγραμμα να λειτουργήσει αν λειτουργήσει. Ευχαριστώ. Thank you. On the first question, no, Σε ευχαριστώ για το, την πρώτη σας ερώτηση. Δεν υπάρχουν δύο διαφορετικές κατηγορίες. Όλες οι τράπεζες υπόκεινται στην ίδια εποπτεία από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. <clears throat> Και από το SSM. Τώρα, η διαφορά μεταξύ των τραπεζών σε σχέση με τις τράπεζες που βρίσκονται στον κατάλογο και εκείνων που δεν βρίσκονται στον κατάλογο είναι η εφαρμογή. Είναι λοιπόν ο βαθμός κεντροποίησης κεντρικού χαρακτήρα και άμεσης λογοδότησης προς το κέντρο. Όμως καταρχήν το σύστημα θα εφαρμόζεται, θα ισχύει για να διασφαλίζει ένα ισοδίκαιο πεδίο δραστηριοποίησης σε όλες τις τράπεζες στον χώρο του ευρώ. Η εφαρμογή υλοποίηση για τις μικρότερες τράπεζες ε, θα απαιτεί μεγαλύτερη συμμετοχή των εθνικών αρμόδιων αρχών σύμφωνα με μια κεντροποιημένη διαδικασία κανόνων κανονισμών. Δεν θα υπάρχουν λοιπόν δύο κατηγορίες. Για το ESM ας αναφερθώ στο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ της 15ης Νοεμβρίου αν επιτρέπετε. Εκεί αναφέρεται ρητά ότι πρώτα απ' όλα έχουμε την ιδιωτική πηγή χρηματοδότησης. Δεύτερον, έχουμε τις εθνικές δυνατότητες χρηματοδότησης. Αν δεν επαρκούν, έχουμε τα μέσα στον χώρο ευρώ, ώστε ο χώρος ευρώ και της, Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιηθεί όπως πρέπει. Πρώτα, η ESM ε θα δώσει μέσω των κανονικών διαδικασιών χρηματοοικονομική υποστήριξη για την ανακεφαλοποίηση των Ιδρυμάτων μέσω δανείων στα κράτη-μέλη, με τον τρόπο που έγινε στην Ισπανία αυτό ακριβώς. Δεύτερον, η άμεση ανακεφαλοποίηση και τα μέσα ανακεφαλοποίηση με 60 δις όσον αφορά το βαθμό έκθεσης στους κινδύνους θα μπορούσε να προσαρμοστεί όσον αφορά τις εθνικές διαδικασίες και κανόνες με τον, ε, τη συμφωνία του, ε, της 30 Ιουνίου μετά από την έγκριση ε, δημιουργίας του ESM. Αυτά είναι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ της 15ης ε, Νοεμβρίου. Τώρα, για το τρίτο σημείο ως παρατήρηση που αναφέρατε, για την δημοσιονομική λιτότητα. Πρώτα απ' όλα, δεν θα έπρεπε να ξεχνάμε βέβαια ποια ήταν η κατάσταση όταν ξεκινήσαμε, όταν τα πρώτα προγράμματα καταρτίστηκαν και σχεδιάστηκαν. Ήταν μια κατάσταση με μεγάλη αβεβαιότητα και ανασφάλεια, δραματικού χαρακτήρα αβεβαιότητα και ανασφάλεια, με σπρέτς των κρατικών ομολόγων, αρκετά αρκετές εκατοντάδες ε, σημεία ανώτερα από ό,τι σήμερα που στραγγάλιζαν ασφικτικά την οικονομία. Είχαμε και την ύφεση. Η πραγματική ύφεση ξεκίνησε λοιπόν τότε σε εκείνη τη φάση. Τα προγράμματα λοιπόν παίρνουν σάρκα και μορφή και οστά σε εκείνη την περίοδο χρονικά. Τότε στο παρελθόν. Και ειλικρινά αν δούμε το τι συνέβη ακριβώς για παράδειγμα στην Πορτογαλία όπου κάποιους μήνες πριν το πρόγραμμα φαινόταν ότι δεν έβαινε καλώς και κάποιες αβεβαιότητες που υπήρχαν λόγω ε, τοποθετήσεων των δικαστηρίων, αποφάσεων δικαστηρίων. Άμεσα οι αγορές ε, ε, έθεσαν κυρώσεις, δημιούργησαν κυρώσεις για την Πορτογαλία και τα ομόλογα. Να πει κανείς ότι ο τρόπος που καταρτίστηκαν και σχεδιάστηκαν αυτά ότι πιθανώς μπορεί να μην ήταν σωστά τότε για εκείνη τη χρονική στιγμή έστω. Αλλά τι θα κάνουμε τώρα για την ε, ε, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μην ανατρέψουμε την πρόοδο που συνέβη και σημειώθηκε και να μην υπονομεύσουμε αυτή την πρόοδο που έγινε μέχρι σήμερα. Να προσαρμοστεί η δημοσιονομική προσαρμογή ώστε να είναι πιο φιλική προς την ανάπτυξη. Δημοσιονομική λοιπόν σταθεροποίηση με μεγαλύτερες κρατικές δαπάνες ε, για τις υποδομές, κεφαλαϊκές υποδομές, να έχουμε λοιπόν και χαμηλότερα επίπεδα φορολογίας και τέταρτον ή τρίτον, τρίτον να κάνουμε, να προβούμε σε διαθροτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις γιατί αυτές είναι οι μόνες που μπορούν να προκαλέσουν και να δημιουργήσουν ανάπτυξη αηφόρα και μακροπρόθεσμα. Με ένα μάθημα μπορούμε να συναγάγουμε και το έχουμε ε, επανειλημμένα δεν είναι δυνατόν με σταθερή και μόνιμη δημιουργία χρέους να υπάρχει αηφόρος ανάπτυξη. Και έτσι δεν μπορεί να υπάρξει ισοδίκαια, ας το πω έτσι, διαδικασία μέσω της δημιουργίας 200 νέου χρέους. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε. από τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να επανέλθω στην κατάσταση που επικρατεί στις χώρες που συνεχίζουν να έχουν δυσκολίες. Αναφερθήκατε στην ανάγκη εφαρμογής μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών σε χώρες όπως είναι η Ιταλία και η Γαλλία για παράδειγμα. Προς το παρόν όμως δεν έχουν γίνει αρκετά πράγματα. Δεν έχουν γίνει πολλά. Ούτε εσείς, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, δεν μπορείτε να επηρεάσετε ώστε οι χώρες αυτές να κάνουν κάτι. Το μόνο που κάνει τις χώρες να αντιδράσουν είναι, όπως είδαμε και με τον ε, Μπερλουσκόνη, όταν ξαφνικά τα επιτόκια ε, ανέβηκαν τόσο πολύ, τότε μόνο αντέδρασε. Ε, εντάξει, τρεις μέρες, τρεις μέρες, γιατί μετά βέβαια σταμάτησε. Έπρεπε να φύγει μετά. Τελείωσε, όσο εκεί ήταν. Αλλά η ερώτησή μου είναι εξή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που ακολουθεί μέχρι τώρα, που προσφέρει δηλαδή στις τράπεζες χρήματα με χαμηλά επιτόκια, φτηνό χρήμα και που έχουν χρησιμοποιήσει στην Ιταλία αλλά και σε άλλες χώρες για να αγοράσουν ομόλογα. Μήπως είναι αντιπαραγωγική με τέτοια πολιτική. Γιατί τότε οι δυνάμεις της αγοράς θα είχαν κατά πάσα πιθανότητα πιέσει τόσο πολύ την κυβέρνηση που τελικά θα είχαν αντιδράσει διαφορετικά. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, κάποιος από τους ε, υψηλά εστάμενους, ο Άσμου Σένο, ο διευθυντής σας, ανακοίνωσε ότι φεύγει. Δεν είμαι από την πολιτική του ομάδα, αλλά λυπούμε γι' αυτό, γιατί είχα την εντύπωση ότι ήταν αποτελεσματικός στην ομάδα σας. Και βλέποντας απ' έξω τα πράγματα, είχα την αίσθηση ότι τα πηγαίνατε και καλά μεταξύ σας. Πολύ καλά μάλιστα θα έλεγα. Οπότε η ερώτησή μου είναι η αναχώρησή του, και εντάξει δεν ψάχνω να βρω τώρα τους λόγους, όποιοι και είναι αυτοί, αλλά ρωτάω, το γεγονός ότι αποχωρεί, τι επιπτώσεις θα έχει στο τμήμα του. Θα οδηγήσει σε κάποια αναδιοργάνωση των αρμοδιοτήτων μεταξύ των διευθυντών. Πλεονέκτημα να, εδώ ο φίλος μου, εδώ εξ αριστερών, θα χαρεί πολύ άμα σας πω να είναι γυναίκα αυτή που θα τον αντικαταστήσει. Και ολόκληρο το Κοινοβούλιο θα χαρεί πολύ αν συμβεί αυτό. Τέλος. Ο Άσμουσεν ήταν κάποιος ο οποίος έθεσε το θέμα κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει ή όχι να δημοσιεύει τα πρακτικά της. Ήταν από τους πρώτους που το έθεσε. Και η συζήτηση έγινε και συνεχίστηκε για πολύ καιρό. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η πολιτική σας όσον αφορά τη δημοσίευση των πρακτικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για την πρώτη ερώτηση, για την πρώτη ερώτησή σας θέλω να απαντήσω το εξής. Κατά πόσο δηλαδή η πολιτική μας ε, είχε σαν αποτέλεσμα να μειωθούν τα κίνητρα των κυβερνήσεων για να αντιδράσουν. Είναι ένα θέμα που έχει τεθεί πολλές φορές μέχρι τώρα. Κοιτάξτε, είναι το αντίθετο. Όταν εμείς δρούμε και νομίζω ότι είναι γνωστό τη σπάση. Υπήρχαν κίνδυνοι με το ευρώ και φημισμό, μάλιστα θα έλεγα ότι υπήρξε δηλαδή μεγάλο σκεπτικισμός για το κατά πόσο το ευρώ θα μπορούσε να επιβιώσει τελικά ή όχι όταν ξεκίνησε το πρόβλημα. Εμεί, πιστεύω ότι αντιδράσαμε και αντιμετωπίσαμε θετικά την κατάσταση με θετικά αποτελέσματα. Αν τώρα δείτε τα επιτόκια των αγορών σε σχέση με τα κίνητρα για μεταρρυθμίσεις, εδώ πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Πιστεύετε ότι μια χώρα θα άλλαζε τον εκλογικό της νόμο, για παράδειγμα, επειδή τα επιτόκια είναι εκατοντάδες μονάδες παραπάνω Πως θα πρέπει. Πιστεύετε ότι μια χώρα θα άλλαζε το εκπαιδευτικό της σύστημα ή το δικαστικό της σύστημα επειδή τα επιτόκια είναι ψηλά, τα επιτόκια δανεισμού. Όχι. Αυτό που θα μπορούσε να κάνει μια χώρα να αλλάξει είναι στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τη δημοσιονομική διαδικασία. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η λιτότητα, οι αποταμιεύσεις θα ακολουθούσαν. Αλλά οι πραγματικές ε, μεταρρυθμίσεις δεν θα τις έκανε μια χώρα, δεν θα άλλαζε την εργασιακή της ας πούμε νομοθεσία εξαιτία των επιτοκίων μια χώρα. Μάλλον όχι. Την έχουμε υπόψη μας λοιπόν αυτή την ε, διάσταση. Είμαστε ευαίσθητοι γιατί θέλουμε να πετύχουμε οι χώρες να υιοθετήσουν τέτοιες μεταρρυθμίσεις. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε την εντύπωση ότι η γενική αβεβαιότητα, αυτή η δραματική αβεβαιότητα που κυριαρχούσε στην ε, Ευρωζώνη θα έχει σαν αποτέλεσμα να αλλάξουν τα πράγματα. Βέβαια έκτοτε κοιτάμε τις χώρες που πρέπει έτσι καλώς να κάνουμε τα ρυθμίσεις, γιατί δεν υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη αν δεν υπάρξουν τέτοιες μεταρρυθμίσεις. Και αν ήταν λιγότερο, δεν σημαίνει ότι χωρίς μεταρρυθμίσεις θα είχαμε ανάπτυξη ακόμα και αν τα επιτόκια δηλαδή δεν ήταν τόσο ψηλά. Τώρα, η αποχώρηση του Γέργα. Είναι μια μεγάλη απώλεια για το Συμβουλίο μας και για μένα προσωπικά. Εσείς είπατε ότι τα πηγαίναμε πολύ καλά, τα πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά εγώ θα έλεγα εγώ. Πολύτιμο συνεργάτης για μένα. Το ξέρω 15 με 20 χρόνια είχαμε φιλία αδερφική και η συνεισφορά του στο έργο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, ήταν κάτι το πολύτιμο, ανεκτήμητη η βοήθειά του. Φυσικά και του εύχομαι ότι καλύτερο για τη συνέχεια. Θα μας λείψει όμως, θα μας λείψει πολύ. Το μόνο που μπορώ να πω τώρα είναι ότι ο αντικαταστάτης του πρέπει να βρεθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα. Πρέπει να υπάρξει μια πολύ γρήγορη αντίδραση από το Συμβούλιο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βέβαια. Πολύ γρήγορα, γιατί πρέπει να συμπληρωθεί και να πληρωθεί η θέση αυτή τη στιγμή που ασχολούμαστε με πάρα πολλά πράγματα. Γιατί είναι και η οικονομική βέβαια πολιτική και η προετοιμασία του ενιαίου οπτικού μηχανισμού κλπ. κλπ. Είναι δηλαδή μια στιγμή που δεν αντέχουμε με ένα τέτοιο κενό, να μας λείπει δηλαδή ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο Γιάρκ ήταν ένας από αυτούς που άρχισε τη συζήτηση για το θέμα της δημοσίευσης των πρακτικών. Είναι κάποιοι όπως και εγώ που νοιαζόμαστε για αυτό το θέμα. Δεν είναι όμως εύκολο. Θέλουμε, γι' αυτό λέω ότι η συζήτηση είναι πιο περίπλοκη από ό,τι περιμέναμε, γιατί πρέπει να ζυγίσουμε από τη μια μεριά την επιθυμία να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Υπάρχει μεγάλη διαφάνεια, να το συγκρίνουμε με τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες, αλλά μας ενδιαφέρει να είμαστε να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλά συγχρόνως να υπάρχει και εθνική ανεξαρτησία των μελών του Δικητικού Συμβουλίου. Δεν θέλουμε δηλαδή τα μέλη αυτά να βρεθούν ε, υποπίεση από τις χώρες τους για να ψηφίζουν βάσει των συμφερόντων της χώρας τους και όχι της, Ευ... της Ευρώπης στο σύνολό της. Σας ευχαριστώ. Είμαστε κάπως απίθαρχοι με τις ερωτήσεις στον χρόνο αυτό βάλουμε τάξη. Για τους συντηρητικού και μεταρρυθμιστές σε σχέτεση τον λόγο κύριε Πίτερ Φαντάρα. Ευχαριστώ πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήσει έχω. Πρώτον, η χώρα μας πιστεύει ότι και ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να μειώσει τα χρέη του γιατί αλλιώ υπάρχει ο κίνδυνος του πληθωρισμού. Και θέλω λοιπόν να ρωτήσω τι μηχανισμούς έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τι μηχανισμούς θα χρησιμοποιήσει για να το πετύχει αυτό. Οι τράπεζες δανείζονται φτηνό χρήμα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έχουμε τα μη συμβατικά μέσα, τις πολιτικές αυτές, τις μη συμβατικές, οπότε η ερώτησή μου είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα από ποια ακόμα ε, χώρα θα αγοράσει ομόλογα, ποια θα είναι η επόμενη χώρα. Έπειτα η Spiegel, ο Σπίγκελ δημοσίευσε ένα άρθρο σχετικά με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με τα ομόλογα της Ιταλίας. Τα κρατικά ομόλογα της Ιταλίας. Το οποίο τα αγοράζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με μια βάση DBRS. Τι είναι? Θέλω να ξέρω. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα υπερτιμήσει τα ομόλογα αυτά. Το Spiegel συνεχίζει με τα DBRS Το άρθρο αυτό δηλαδή αναρωτιέται για την ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οπότε θέλω να ξέρω κι εγώ γιατί αναμειγνύει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γιατί θα πρέπει να δοθεί και κάποια απάντηση στο δημοσιογράφο. Uh, let me, ε, let me clear... Να είμαι ξεκάθαρος για... Να αμέσως τη δεύτερη ερώτηση. Τότε δεν είχαμε διαφορετική εφαρμογή έναντι άλλη περίπτωση. Δεν χρησιμοποιήθηκε κάποιο ειδικό μέτρο για την Ιταλία ή άλλη χώρα. Αυτή είναι η κανόνε Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και τελεία και παύλα. Για το πρώτο σημείο που αναφέρατε <clears throat> για την ε, deflation, δεν βλέπουμε λοιπόν στασιμό πληθωρισμό με τον όρο και ορισμό δηλαδή να υπάρχει και μείωση και τιμών όπου αναβάλουν τα προγράμματα δαπανών τους οι πολίτες επειδή πιστεύουν ότι κάποτε θα μειωθούν οι τιμές και γι' αυτό κάποτε όταν θα έπεφταν θα αγόραζαν. Δεν βλέπουμε τέτοια κίνηση. Δεν βλέπουμε μια γενικευμένη μείωση τιμών όσον αφορά αγαθά στις ε, χώρες μας. Δεν βλέπουμε μια κατάσταση όπως στην Ιαπωνία με το στασιμοπληθωρισμό όπου η κύρια διαφορά σε σχέση με το ερώτημα βρισκόμαστε εμείς σε μια παρόμοια κατάσταση με την Ιαπωνία και βλέπουμε τις διαφορές. Οι διαφορές είναι ουσιαστικά ότι μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οι προσδοκίες ε, για τον πληθωρισμό είναι καθορισμένες. Ε, σε σχέση με την Ιαπωνία δεν ήταν, σε σχέση με τη δεκαετία 90, αρχές ε, το, της δεκαετίας του 2000. Αυτό είναι ένας λόγος. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα νομισματικά κίνητρα στη δική μας περίπτωση ήταν πολύ ισχυρότερα από εκείνα τα κίνητρα στην Ιαπωνία τότε στο παρελθόν και ο τρίτος λόγος είναι ότι ειλικρινά η κατάσταση των τραπεζών και του ιδιωτικού τομέα στην Ιαπωνία κατά τα τέλη της, όταν έσπασε η φούσκα των ακινήτων κατά τα τέλη της δεκαετίας του 80 αρχές της δεκαετίας του 90 ήταν πολύ χειρότερη η κατάσταση από ότι σήμερα στην Ευρώπη η κατάσταση. Και ο τέταρτος λόγος, ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους είναι ότι ουσιαστικά εμείς ξεκινάμε με τις δοκιμές ε, για τις τράπεζες ε, στο σύστημά μας πολύ πρόωρα και έγκαιρα, πολύ νωρίς, πράγμα το οποίο δεν συνέβη στην Ιαπωνία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα έπρεπε λοιπόν να θυμόμαστε ένα πράγμα πάντα. Η νομισματική πολιτική για να έχει αποτελέσματα στις τιμές ε, και στις επιδόσεις πρέπει να διαβιβάζεται και να περνάει στους πολίτες και χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα. Παίρνει κάποιο χρονικό διάστημα προτού μπορέσει να περάσει στην πραγματική οικονομία το μήνυμα και τα κίνητρα της νομισματικής μας πολιτικής. Τώρα η ταχύτητα διαβίβασης της νομισματικής μας πολιτικής εξαρτάται από το πόσο υγιές είναι το τραπεζικό σύστημα. Όσο υγιέστερο είναι το ε, τραπεζικό σύστημα τόσο ταχύτερη θα είναι η μεταβίβαση. Αυτή είναι μία άλλη σύγκριση με την κατάσταση της Ιαπωνίας κατά το παρελθόν. Και γι' αυτό από πλευρά EQR ε, θα έχουμε επιτάχυνση της ε, ταχύτητας ε, μεταβίβασης ή διαβίβασης μεταξύ δηλαδή των κινήτρων και του αποτελέσματος που θα επιτευχθεί στην πραγματική οικονομία. Από την άλλη πλευρά έχουμε πολλά μέσα και εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε το στασιμό πληθωρισμό. Δεν βλέπουμε τέτοιο κίνδυνο να υφίσταται σήμερα. Όμως έχουμε συνειδητοποιήσει απόλυτα και πολύ καλά ότι για να τηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα ο πληθωρισμός πολύ κάτω από το 2% όριο για μακρόχρονικό διάστημα έχει κινδύνους που συνεπάγεται αυτή η πολιτική και είμαστε πρόθυμοι και έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και να δράσουμε σε, αυτή τη, σε αυτό το μέτωπο. Την Γκόρτ από τους Πρασίνους παρακαλώ. Ευχαριστώ και καλώς ήρθατε πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ανάμεσά μας. Δύο γρήγορες γοργές ερωτήσεις. Για το τι συνέβη με τον κύριο Άσμουσεν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι με την αποχώρησή του θα χάσετε ένα ε, σου άτομο. Κάποιον δηλαδή που στο κοινό στους Γερμανούς πολίτες ήταν υπέρ του προγράμματος που είχε ξεκινήσει. Και παρόλη αυτή την υπεράσπιση η εικόνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Γερμανία υπέστη μια ευθύνουσα πορεία και τάση κατά το τελευταίο διάστημα στη Γερμανία. Ποια είναι η στρατηγική για να πληρωθεί αυτό το κενό του κυρίου Άσμουσεν. Γιατί ένα πράγμα ήδη το βλέπουμε. Θα είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει ένας, μια γυναίκα ε, πραγματικά καταρτισμένη και ικανή ε, και επιδέξια στο πλευρό σας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που θα αναπληρώνει τον κύριο Άσμουσεν. Θα ήθελα δεύτερο να μου πείτε πώς είπατε παρακαλώ. Μα πραγματικά δημονώ να δω ότι θα συμβεί τώρα. Στα γερμανικά συνεχίζει ο μιλητής. Αδειμονώ να δω τι θα συμβεί. Πέρα από όλα αυτά θα ήθελα να μου πείτε όσον αφορά το SRM θα μπορούσατε να είσαστε πιο επακριβείς και εξειδικευμένο στην τοποθέτησή σας. Σε ποιο βαθμό σε σχέση με το κείμενο του Συμβουλίου δεν υπάρχει ανταπόκριση σε μια πραγματικά ευρωπαϊκή και ένα αποτελεσματικό ευρωπαϊκού χαρακτήρα μέσο το οποίο απαιτούσατε και ζητούσατε. Yeah. Εσείς τώρα Τελευταίος αγορητής παρακαλώ. Θα έλεγα ότι όπως προαναφέρθηκε λέει ο κύριος Ντράγκη θα μας λείψει πραγματικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ο κύριος Άσμουσεν. Θα είναι πολύ αισθητή η απουσία του. Και αυτό το οποίο αναφέρθηκε για την νομισματική πολιτική για το σύνολο της ζώνης ευρώ. Τώρα ανα, αναγνωρίζεται πάρα πολύ από όλους ότι ήταν ένα πολύ επιτυχημένο μέτωτο Και λυπούμε ότι στη Γερμανία κάποιοι μπορεί να μην συμφωνούν με αυτό το γεγονός. Όμως παγκόσμια αναγνωρίζεται ότι είχε στεφθεί και με επιτυχία. Πραγματικά εύχομαι, θα ευχόμουν ε, εκείνος ή εκείνη που θα διαδεχθεί τον κύριο Άσμουσεν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα έχει όλες τις αρετές και όλες τις ικανότητες που έχει ο κύριος Άσμουσεν. Ίσως και περισσότερες ακόμα. Εξαρτάται από το πώς εκείνος ή εκείνη θα ε, δρα, ε, δραχθεί της ευκαιρίας και θα δραστηριοποιηθεί και ποια καθήκοντα θα αναλάβει. Δεν είναι δικό μου έργο να επιλέξω εγώ την ή τον διάδοχο του κυρίου Άσμουσεν. Είναι θέμα του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο γνωρίζει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι πρέπει να είναι ικανός, ικανό άτομο ο διάδοχος του Άσμουσεν. Ικανό επαγγελματικά με υψηλού επίπεδου ε, ικανότητες και γνώσεις και πρέπει γοργά να αναπληρωθεί αυτό το κενό. Αυτό είναι χέρια σημασίας. Πρέπει γοργά να αναπληρωθεί το κενό που θα προκαλέσει η απουσία του κυρίου Άσμουσεν. Αν γίνει γοργά λοιπόν αυτό και αναπληρωθεί γοργά, τότε το πρόβλημα της απουσίας του κυρίου Άσμουσεν σύντομα θα επιληθεί και θα είναι πλήρες σε απαρτία το Συμβούλιο και θα είναι σε θέση πλέον να αντιμετωπίσει τις πάμπολες προκλήσεις που θα αντιμετωπίζουμε στο μέλλον. Τώρα, για το ε, SRM, η έννοια να έχουμε μία αρχή, μία προσέγγιση ενιαία και ένα ταμείο είναι ακριβώς η προσέγγιση που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τα πράγματα βαίνουν καλώς λοιπόν ως προς αυτό αν ακολουθηθεί αυτή η πορεία. Υπάρχει όμως και μια άλλη πτύχη όπου εμείς θα επιθυμούσαμε να βλέπαμε οι δύο, τις δύο φάσεις αυτής της διεργασίας να είναι σαφώς διαχωρισμένες να διαχωριστούν. Θα έπρεπε η αξιολόγηση από την ε, ε, επιτήρηση, εποπτεία για τη μη βιωσιμότητα κάποιων τραπεζών θα πρέπει να διαχωρίζεται σαφώς από τις αποφάσεις του SRM, του τι θα πρέπει να γίνει για αυτές τις μη βιώσιμες τράπεζες. Τώρα, σήμερα, υπάρχει κάποια σύγχυση ή ένα σύμφυρμα αρμοδιοτήτων, όπου το SRM θα μπορούσε να έχει κάποιο λόγο να αρθρώσει στη μη βιωσιμότητα κάποιας τράπεζας. Όταν αυτά τα πράγματα γίνονται με σωστό, σωστό τρόπο, τα δύο πράγματα αυτά πρέπει να διαχωρίζονται και διαχωρίζονται απόλυτα. Γιατί οποιαδήποτε αρχή που θα αξιολογεί θα πρέπει να έχει και κάποια δυνατότητα να ε, δούμε πώς μπορεί να παραταθεί ή να επεκταθεί αυτή η διαδικασία. Θα πρέπει να γνωρίζουν όμως ε, ένα πράγμα. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να είναι χρονοβόρα. Πρέπει να γίνονται άμεσα. Υπάρχει ένα σημείο μη βιωσιμότητας. Όταν διατυπώνει κάποιος επιτηρητής επόπτης ότι κάποιο θεσμικό όργανο κάποια τράπεζα δεν είναι βιώσιμη, τότε οποιαδήποτε συναλλαγή ή οποιαδήποτε κίνηση μπορεί να εντάσσεται υπό την διαδικασία του ε, δικαίου ε, για την πτώχευση ή χρεοκοπία. Πρέπει άμεσα να λαμβάνονται αποφάσεις, διότι μπορεί κάποιες τράπεζες να μην είναι βιώσιμες, αλλά δεν πρέπει να αναφέρεται αυτό ότι δεν είναι βιώσιμες. Διαφορετικά θα δημιουργηθεί μια χαόδης κατάσταση που θα πρέπει να διαχειριστούμε κατά το άμεσο μέλλον. Γι' αυτό οποιοδήποτε μηχανισμός θεσπιστεί για να λειτουργήσει θα πρέπει να λειτουργεί άμεσα. Όχι να έχουμε εκατοντάδες άτομα που θα διαβουλεύονται αν κάποια τράπεζα είναι βιώσιμη ή όχι και θα παρατείνονται οι διεργασίες. Αυτή είναι η ανησυχία μου. Ο μηχανισμός που θα δημιουργηθεί να είναι ένας βιώσιμος, λειτουργικός, αποτελεσματικός μηχανισμός. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, η ερώτηση ξεκινάει η ερώτησή μου ξεκινάει από την ελλάδα αλλά νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον για όλη την ευρωπαϊκή ένωση οπωσδήποτε για τον ευρωπαϊκό νότο. στην ελλάδα υπάρχει αυστηρή λιτότητα που επέβαλε η τρόικα είσαστε μέλος της οι μισθοί έχουν μειωθεί πάνω από το 50% έχουν γίνει πολλές μεταρρυθμίσεις στην αγορά υπηρεσιών και εμπορευμάτων για να φύγουν τα εμπόδια αλλά στην ελλάδα υπάρχει πτώση ρεκόρ στις εξαγωγές 12% η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 5%. Η ανεργία έχει πάει στο 30%. Την ίδια στιγμή που τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μειώνονται, το 60% των ελληνικών επιχειρήσεων μείωσαν τις επενδύσεις. Το 25% έχει ρευστότητα. Αποτέλεσμα. Πολλές μεγάλες επιχειρήσεις, κύριε Πρόεδρε, φεύγουν από την Ελλάδα και από τον Νότο ενδεχομένως και κατευθύνονται στη βόρεια ευρώπη για να βρουν φθηνότερο δανεισμό. στο νότο τα επιτόκια μειώνονται αυξάνονται συγγνώμη, με συνέπεια να πνίγουν οικοκυριά και επιχειρηματικότητα ενώ στις βόρειες χώρες στη γερμανία μειώνεται με συνέπεια να συγκεντρώνει τα, όλα τα χρήματα και όλες τις επενδύσεις. ρωτηθήκατε και πριν τα προγράμματα όσο αφορά την ελλάδα για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της τρόικα μέσω των εσπα έχουν αποτύχει. η ερώτηση λοιπόν κύριε πρόεδρε είναι πώς θα φέρετε ισορροπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την οποία μιλάτε. Πώς, τι μέτρα θα πάρετε να σταματήσετε να στρέφονται οι επενδύσεις και οι επιχειρήσεις προς τη Βόρεια Ευρώπη, προς τη Γερμανία, τη στιγμή που ο Νότος βυθίζεται στην ύφεση και την ανεργία. Ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστώ. Η απάντηση στην ερώτησή σας είναι μία και μοναδική. Πρέπει πραγματικά να πολεμήσουμε τον κατακαιρματισμό. Και έχουμε πετύχει πολύ σημαντική πρόοδος προς αυτό σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή στην καταπολέμηση του κατακαιρματισμού όσον αφορά κυρίως την χρηματοδότηση. Οι τράπεζες είναι πλέον σε θέση να χρηματοδοτούνται οι ίδιες σε επιτόκια τα οποία διαφέρουν και έτσι ακριβώ θα πρέπει να είναι, σε σχέση βέβαια με τον κίνδυνο, σε σχέση με τι προποθέσει κινδύνου. Δεν διαφέρουν όμω τα επιτόκια όσο διέφεραν πριν απο έναν χρόνο. Αν μάλιστα συγκρίνουμε τώρα την διασπορά που υπάρχει ανάμεσα στις, στα επιτόκια που πληρώνει οι τράπεζες για να χρηματοδοτηθούν από καταθέσεις, βλέπετε ότι η απόσταση βρίσκεται πάνω κάτω στο επίπεδο που βρισκόταν το 2007. Αν μιλάμε λοιπόν για χρηματοδότηση και αν μιλάμε για χρηματοδότηση μέσω καταθέσεων, ο εν λόγω κατακαιρματισμός έχει εξαφανιστεί. Ωστόσο, οι τράπεζες χρηματοδοτούνται και με άλλους τρόπους, μέσω των ομολόγων, μέσω της έκδοσης ομολόγων. Εκεί συγκεκριμένα βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορές ως προς το κόστος. Σημαντικές διαφορές ακόμα. Τώρα, όσον αφορά την πλευρά της δανειοδότησης, προφανώς υπάρχει ακόμα κατακαιρματισμός. Οι τράπεζες δηλαδή χρεώνουν αυτή τη στιγμή επιτόκια, τα οποία διαφέρουν πολύ ανάμεσα στη Βόρεια και τη Νότια Ευρώπη και οι προποθέσει δανειοδότηση επίση διαφέρουν πολύ από τη μία χώρα στην άλλη, από τη μία περιοχή στην άλλη. Αλλά ακόμα και εκεί βλέπουμε κάποιε βελτιώσει, οι οποίε όμω είναι πολύ πιο μικρέ. Τώρα, βλέπουμε από την άλλη κάτι θετικό και το είπα αυτό και στην αρχική μου τη δήλωση, ότι η ροή της δανειοδότησης, η οποία ναι μένει υποτονική, παρόλα αυτά δεν συνεχίζει να επιδεινώνεται, τουλάχιστον στα τελευταία δεδομένα που έχουμε. Υπάρχει δηλαδή μια πολύ μικρή μείωση, αλλά δεν έχουμε την έντονη αυτή πτωτική τάση που είχαμε στο παρελθόν. Είμαι πεπισμένος ότι καθώς ανακάμπτει σιγά σιγά η οικονομία θα δούμε σιγά σιγά βαθμιαίαν εξαφανίζονται τα προβλήματα αυτά. Ωστόσο δύο βασικά στάδια πρέπει να επιτευχθούν για να καταπολεμήσουμε την, τον κατακαιρματισμό. Να αρχίσει να λειτουργεί καταρχάς ο SSM, ο ενιαίος υποπτικό μηχανισμός. Ας μην ξεχνάμε ότι μια συνιστόσα του κατακαιρματισμού, ένας λόγος κατακαιρματισμού, είναι ότι ξαφνικά είδαμε ότι διαφορετικοί πολίτες σε διαφορετικές περιοχές της Ευρωζώνης άρχισαν τελικά να μην έχουν εμπιστοσύνη στις τράπεζες άλλων περιοχών της Ευρωζώνης. Υπήρχε δηλαδή μια κατάρρευση της ίδιας εμπιστοσύνης στην Ευρωζώνη που ουσιαστικά δημιούργησε πάλι ανόρθωσε κάποια εθνικά σύνορα. Πιστεύω ότι στα πλαίσια του ενιαίου υποπτικού μηχανισμού θα έχουμε πλέον ένα ισότιμο πεδίο εποπτείας στην Ευρωζώνη και αυτό θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε αυτή την έλλειψη εμπιστοσύνης. Ο δεύτερος μηχανισμός βέβαια είναι ο SRM, ο ενιαίος μηχανισμός εξυγίανσης, το ότι θα έχουμε πλέον ενιαίο σύστημα για την εξυγίανση και την ακαθάριση των τραπεζών και αυτό θα επιτελείται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σε όλες τις περιοχές της Ευρωζώνης. Και αυτό αποτελεί πολύ σημαντική συνιστόσα. Τρεις παράγοντες βασικά βλέπουμε, καθώς προχωρά και βελτιώνεται η οικονομία, η αποφυγή του κινδύνου, η οποία είναι υψηλή ακόμα στον Νότο, ουσιαστικά θα μειωθεί. Και ήδη βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει μία πρόοδος ως προς αυτό στις νότιες χώρες και στην Ελλάδα. Πρώτος λόγος αυτός. Δεύτερον, θα αρχίσει να ισχύει πολύ σύντομα ο ενιαίος υποπτικός μηχανισμός και τρίτον θα αρχίσει να ισχύει και ο ενιαίος μηχανισμός εξυγίανσης. Όσο προχωράμε προς μια πραγματική τραπεζική ένωση, όσο περισσότερο διασπάμε το σύνδεσμο ανάμεσα στα κρατικά ομόλογα και τις τράπεζες, τόσο περισσότερο θα είμαστε σε θέση να κερδίσουμε τη μάχη κατά του κατακαιρματισμού. E Ευχαριστώ. Σαν από το EFT. Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ που ήρθατε στην κοινοβουλευτική μας επιτροπή και πάλι κύριε Ντράγκη όπως είπατε πιο πριν, παίρνει χρόνο μέχρι ότου να λειτουργήσουν σωστά οι αποφάσεις μας. Όλοι συμφωνούν ότι με μεγάλη βραδύτητα αντέδρασε στην κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε απλά προετοίμαστοι τότε και δεν αντιδράσαμε έγκαιρα. Λοιπόν, συχνά κάνουμε λόγο για προγραμματισμό και σχεδιασμό λύσεων για υποθετικέ κρίσει στο μέλλον. Όμω ταυτόχρονα πρέπει να επιλύσουμε τα σημερινά επίκαιρα προβλήματα. Ξέρουμε ότι η ελληνική περίπτωση δεν έχει επιλύθει και έχουν εξαντληθεί από τη λιτότητα οι πολίτε σε κάποια κράτη-μέλη. Το μεγαλύτερο ζήτημα και στο ε, κοντινό και στο απότερο μέλλον είναι η δυνατότητα ίσω για κάποια κράτη-μέλη να εξέλθουν, να αποχωρήσουν από τη ζώνη ευρώ. Αυτό ρωτάνε και οι πολίτε και οι ερευνητέ για παράδειγμα, τον προηγούμενο μήνα ο κύριος Φρανκ Νιούμαν που ήταν αναπληρωτής ε, Υπουργός Οικονομικών είπε σε σχέση με τον ε, τύπο στην Φινλανδία ότι πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα εξόδου από, την, ε, από το ευρώ Βλέπετε ότι είναι εύθετο να έχει προγράμματα η Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχει προγράμματα να είναι προετοιμασμένη για μια τέτοια αποχώρηση κράτους μέλους από το ευρώ, αν αποφασίσει κάποιο κράτος μέλος να αποχωρήσει από τη ζώνη ευρώ, ώστε να μην είμαστε απροετοίμαστοι στο μέλλον. Συζητείτε αυτό το θέμα και στα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να συμμετάσχουμε στη συζήτηση και να προετοιμαστούμε διότι θα ήταν καλύτερη ίσως η κατάσταση σήμερα που ίσως δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για κάτι τέτοιο και η συζήτηση αυτή δεν θα πρέπει να διαδώσει, να μεταδώσει πανικό. Ευχαριστώ. Thank you. I can give you one short... Ευχαριστώ μια ε, συντομότερη και μια μακρότερη απάντηση, μακρύτερη απάντηση, η σύντομη απάντηση. Δεν βλέπω κάποιο κέρδος στο να έχουμε σχέδια αναδίπλωσης ε, το ευρώ, η πορεία στο ευρώ και η κατάσταση με το ευρώ είναι κάτι αμετάκλητο. Δεν είναι κάποια εναλλακτική λύση, είναι κάτι αμετάκλητο. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και τώρα, η κάπως μακρύτερη απάντηση είναι η εξής και αυτό αληθεύει για όλες τις χώρες ουσιαστικά. Ακόμα και με μια πεφωτισμένη ανάλυση το τι θα μπορούσε κάποιος να κερδίσει από μια έξοδο. Αυτά όλα είναι εφήμερα σενάρια. Αν χώρες αποχωρήσουν από το ευρώ επειδή μπορούν να πιστέψουν ότι θα αποφύγουν διαθροτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις θα είναι λανθασμένο. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να κάνουν αυτές τις αλλαγές και μεταρρυθμίσεις εκτός ευρώ και οι συνολικοί όροι και προϋποθέσεις θα ήταν πολύ δυσχερέστερες και πολύ πιο θα έλεγα δύσβατες εκτός ευρώ. Επίσης υπάρχει και μια αφελής προοπτική όπως ε, ακούγεται καμιά φορά πόσο ωραίο θα ήταν να φεύγαμε από το ευρώ και να είχαμε υποτίμηση νομίσματος κατά 40%. Και με το μαγικό ραβδί νομίζουν ότι όλα αυτά θα επιληθούν. πιστεύουν ότι όλα θα, ήταν, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σωστά με μια υποτίμηση 40% ενός νομίσματος χωρίς να υπάρξει καμία διαθωτική αλλαγή από πλευράς αυτών των χωρών. απίθανο και απίστευτο φαίνεται αυτό. Για το ΕΛΚ τώρα έχετε εσείς τον λόγο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ και πρέπει να πω εδώ ότι έχουμε συζητήσει πολλά από τα θέματα με τον κύριο Ντράγκη. Ένα ερώτημα σε σχέση με εσάς κύριε Ντράγκη θα, θα είχα και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που αναφέρεται ότι έχει διαδραματίσει και διαδραματίζει μείζωνα ρόλο για την αντιμετώπιση της κρίσης. Κάτω Σεπτέμβριο στη Ρώμη έγινε μία σύνοδος ε, όπου ε, δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, κ. Ντράγκη ότι μεσοπρόθεσμα η νομισματική σταθερότητα θα πρέπει να είναι το επίκεντρο των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και κάνει και ένα σχόλιο ότι στο α, μέλλον ή και στο παρόν ίσως θα έχουμε περισσότερες δυνατότητες από ό,τι είχαμε, θα είχαμε το παρελθόν. Θα μπορούσατε να σχολιάσετε με περισσότερες λεπτομέρειες ποιες είναι αυτά, ποια είναι αυτά τα μέσα, αυτά τα πρόσθετα μέσα και εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας από πλευράς Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα έτσι. Ευχαριστώ. Well, the, um, the οι τελευταίες μακροοικονομικές προβολές που είχαμε αρχές Δεκεμβρίου δείχνουν ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει χαμηλά στο επίπεδο του 2% μεσοπρόθεσμα. Μεσοπρόθεσμα είναι η πρόβλεψη που χρησιμοποιούμε στον καθορισμό του στόχου μας για τον πληθωρισμό. Συνήθως πηγαίνουμε πέρα από τα δύο χρόνια. Πάντω για το 2014 και το 2015 ο πληθωρισμός θα παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα. Βλέπουμε κάποιου κινδύνους πληθωριστικού εξαιτία των τιμών των πρώτων υλών, ενέργεια, τροφίμων κλπ. Αλλά πρέπει να πω εδώ ότι το χαμηλό επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας θα ε, παρέμβει και αυτός. Οπότε θα κρατηθεί χαμηλό πληθωρισμός. Αν δούμε για τα τρόφιμα και την ενέργεια τον πυρήνα του πληθωρισμού, θα δούμε ότι είναι υψηλότερος από τον συνολικό πληθωρισμό. Αυτό σημαίνει ότι το χαμηλό κομμάτι του πληθωρισμού εξαρτάται από την ενέργεια, τα τρόφιμα και άλλα αγαθά, πώς προβάλλεται δηλαδή για τα επόμενα χρόνια ο πληθωρισμός αυτά. Τα χαμηλά επίπεδα πάντως πληθωρισμού σημαίνει ότι μπορεί να πάει και ακόμα πιο χαμηλά. Αυτό είναι ο κίνδυνο. κάτι το οποίο δεν μα αρέσει, δεν το θέλουμε, γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διάφορα προβλήματα. Ένας λόγος που οι προκάτοχοί μας αποφάσισαν ότι το 2% είναι το σωστό νούμερο, ήταν ακριβώς ότι μπορεί, αν πάει πολύ χαμηλό πληθωρισμός, να πάει κάτι στραβά. Οπότε 0,6% ναι, αλλά μπορεί να είμαστε ήδη σε αποπληθωρισμό εξαιτίας κάποιων σφαλμάτων σε ορισμένε χώρε. Γι' αυτό λοιπόν εμεί θέλουμε το επίπεδο του πληθωρισμού να μένει κοντά, αλλά πάντα κάτω από το 2%. Καταλαβαίνω ότι οι χώρε πρέπει να ξαναδούν τι τιμέ του. Ξέρω ορισμένε χώρε που είναι χρεωμένες που προσπαθούν να αυξήσουν τους τρέχοντες ε, λογαριασμούς τους, να βελτιώσουν τις ανισορροπίες. Γίνεται αυτό και αυτό αποτελεί πρόοδο. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να ξαναδούνε και τις τιμές των εξαγωγών και των εισαγωγών. Κάτι το οποίο είναι πιο εύκολο αν υπάρχει ένας πληθωρισμός κοντά στο 2% από ότι αν έχετε μηδέν πληθωρισμό εξαιτίας της ονομαστικής ε, ακαμψίας που διαπιστώνεται. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι ελοχεύει αυτός ο κίνδυνος και έχουμε μηχανισμούς για να τον αποφύγουμε. Είπαμε ότι προς το παρόν όλα τα επιτόκια, όχι μόνο της αναχρηματοδότησης, όλα τα επιτόκια θα μείνουν επί του παρόντος σε χαμηλό επίπεδο για αρκετό χρονικό διάστημα. Δεν έχουμε την αίσθηση δηλαδή ότι μας λείπουν τα μέσα να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Συνεχίζουμε βέβαια να εξετάζουμε τι άλλα μέσα μπορούμε να έχουμε αν υλοποιηθούν παρετέρω κίνδυνοι. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, πάλι εκ μέρους του ΕΛΚ. Ο κύριος Βέρνερ Λάγκεν, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Προ τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τρει ερωτήσει έχω. Η πρώτη αφορά συνέντευξη που δώσατε σε μια γαλλική κυριακάτικη εφημερίδα όπου ζητήσατε από την κυβέρνηση τη Γαλλία να προβεί σε μεταρρυθμίσει. Κρούσατε κόδωνα κινδύνου. Τίθεται το ερώτημα. Είναι ο στενότερο τομέα αρμοδιοτήτων αυτό τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή τον ξεπερνάτε τον τομέα αυτή η παρέμβασή σα. Ξέρουμε υπό την ιδιότητά σα ω Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Διακόπτει ο μιλητής. Βένερ μπορείς να ξαναξεκινήσεις. Νομίζω θα έπρεπε να τα ξαναπείς. Εντάξει, ευχαρίστως. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, τη γαλλική κυβέρνηση και τον Γάλλο πρόεδρο κύριο Ολάν καλέσατε και την καλέσατε να προβεί σε μεταρρυθμίσει το Σαββατοκύριακο σε μια συνέντευξη τύπου σε μια εφημερίδα. Ερώτησή μου, πώς βλέπετε το έργο σας σε σχέση με τις εθνικές υποχρεώσεις ε, για μια μεταρρύθμιση, για μια ημερήσια διάταξη για μεταρρυθμίσεις. Μια και με, την απόφαση για την Ιταλία <coughs> δεν ε, ε, πρόκειται να αγοράζονται πλέον, ομόλογα, κρατικά ομόλογα και ε, σε σχέση με τον κύριο Τρισέ υπήρξε και ένα άρθρο το οποίο είχε συνταχθεί. Πώς εκτιμάτε τον ρόλο του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε μια διαδικασία μεταρρυθμίσεων όταν υπάρχουν τέτοιες παρεμβάσεις. Δεύτερο ερώτημα, το, η πολιτική του φθηνού χρήματος φθηνό χρήμα. Πώς προβλέπετε και τι προβλέπετε να γίνει σε ευθυγράμμιση με την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ. Όταν εκεί θα επέλθει η καμπή, η αλλαγή, ίσως στην Ιαπωνία όχι ακόμα, αλλά στην, στις ΗΠΑ να αυξηθούν τα επιτόκια. Υπάρχει κάποια διεθνή συμφωνία ή είναι κάτι το απόλυτα ανεξάρτητο και αποσυνδεδεμένο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μια τέτοια λήψη απόφασης. Το τρίτο ερώτημα αφορά τον κύριο Άσμουσεν. Λυπούμε για το ότι αποχώρησε. Αλλά υπήρξε και μια σειρά διαφορών μαζί του. Τουλάχιστον αυτό έλεγε ο τύπο, Και υπήρχαν δημοσιεύματα στον τύπο για τέτοιε διαφορές μαζί του. Συμβαίνει αυτό το οποίο είπατε, ότι ο κύριος Άσμουσεν είναι ο δεύτερος καλύτερος φίλος ε, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τι αληθεύει και τι ισχύει. Να απαντήσω πρώτα στην τελευταία ερώτηση. Είπα ότι η απώλεια του ε, Γιώργα είναι πολύ σημαντική όντως. Και προφανώς είχαμε και έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση. Πρέπει να σας πω όμως ότι ε, η φιλία έχει να κάνει και με τον ε, αμοιβαίο σεβασμό των διαφορετικών απόψεων. Πολλές φορές όντως μπορεί να υπήρχε διάσταση απόψεων ως προς το τι θα πρέπει να γίνει. Αλλά αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό στα πλαίσια των συζητήσεων που έχουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ. Διαφορετικά θα ήμασταν σαν σε ένα σοβιετικό κοινοβούλιο να πρέπει να συμφωνούμε πάντα για τα πάντα. Και προφανώς δεν λειτουργούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημά σας για τις Ηνωμένες όχι, κοιτάξτε. Εμείς ε, οι κεντρικοί τραπεζίτες ουσιαστικά είμαστε πολύ προστατευτικοί αν θέλετε της ανεξαρτησίας μας. Δηλαδή αποφασίζουμε για την νομισματική μας πολιτική βάση της εντολής μας έχει δοθεί, εν προκειμένου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μεσοπρόθεσμη σταθερότητα των τιμών. Ξέρετε ότι στις ΗΠΑ είναι η σταθερότητα των τιμών αλλά και η πλήρης απασχόληση, επιπλέον δηλαδή αρμοδιότητα εκεί εμείς αυτή τη στιγμή δεν συντονίζουμε τις νομισματικές μας πολιτικές. Πριν από πολλά χρόνια, σε ορισμένες περιστάσεις είχαμε ένα κάποιο συντονισμό, ιδίως όσον αφορά τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Αλλά κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Τώρα όσον αφορά το ζήτημα του φθηνού χρήματος. Θα πρέπει να ξέρετε ότι ε, ο ισολογισμός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συρρυκνώνεται πολύ γρηγορότερα από οποιαδήποτε άλλη εθνική κεντρική τράπεζα οπουδήποτε στον κόσμο. Η απάντηση λοιπόν είναι πολύ απλή. Εμείς δεν έχουμε ένα πρόγραμμα εξαγοράς κρατικών ομολόγων όπου αγοράζουμε δισεκατομμύρια κρατικών ομολόγων στην περίπτωση της Κεντρικής Τράπεζας των Πολιτειών υπήρχε όντως ένα πρόγραμμα το οποίο προέβλεπε εξαγορά ενός τρισεκατομμυρίου περίπου ε, ομολόγων σε τήσια βάση. Στην περίπτωση της Ιαπωνίας έχουμε ακόμα πιο θεαματικά δεδομένα και στο Μένο Βασίλειο υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα εξαγοράς κρατικών ομολόγων με συγκεκριμένους αριθμούς. Εμείς δεν έχουμε λοιπόν κάτι τέτοιο. Γι' αυτό το λόγο, στα πλαίσια του δικού του ε, τραπεζικού ισολογισμού γνωρίζουμε ότι η έξοδος από την κρίση είναι ακόμα μακριά, αλλά θα είναι πολύ πιο εύκολη για μας, γιατί ο ισολογισμός μας τελικά ακολουθεί τα LTROs, δηλαδή το πρόγραμμα αναχρηματοδότησής μας. Και όπως σας είπα και στην ομιλία μου, οι τράπεζες ήδη έχουν ξεκινήσει να αποπληρώνουν την πρώτη χρηματοδότηση που τους έδωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα έχει αυτό επιπτώσει τα επιτόκια, δεν νομίζω και δεν θα έπρεπε γιατί η ρευστότητα ουσιαστικά αυτή είναι μια ρευστότητα που ποτέ δεν έγινε πραγματικό χρήμα. Πρόκειται για ρευστότητα η οποία δεν χρησιμοποιήθηκε και επομένω οι τράπεζε είναι σε θέση να την αποπληρώσουν. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λοιπόν βρίσκεται σε καλύτερη θέση σε σχέση με τι άλλε εθνικέ τράπεζε αλλού στον κόσμο. Ωστόσο γνωρίζουμε ότι όντω υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι οι οποίοι προέρχονται από τα χαμηλά επίπεδα πληθωρισμού για ένα παρελθαμένο χρονικό διάστημα. Αυτό το έχουμε πάντα κατά νου. Και κάτι ακόμα, ναι. Αν κατάλαβα καλά, αναφερθήκατε στις εθνικές ευθύνες, εθνικές αρμοδιότητες. Νομίζω ότι οι κυβερνήσεις είναι αυτές οι οποίες είναι τελικά υπεύθυνε στη τελευταία ανάλυση για τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Ωστόσο, υπάρχει κάτι σημαντικό που πρέπει οι κυβερνήσεις να έχουν πάντα κατά νου. Κάτι το οποίο το βλέπουμε όλο και περισσότερο, καθότι συνεργαζόμαστε όλο και περισσότερο με τις εθνικές κυβερνήσεις, όλο και περισσότερο μετά την κρίση. Ένα από τα σημαντικά διδάγματα που αντλήσαμε από την οικονομική κρίση είναι ότι η εθνική πολιτική που ακολουθείται όσον αφορά την οικονομία έχει δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στην Ευρωζώνη. Συνεπώς, υφίσταται ένα κοινό συμφέρον στο να καταρτήσουμε πολιτικές όπου δεν θα έχουμε αρνητικές δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλες χώρες. Άρα πρέπει να αναλυφθούν όλες οι απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, γιατί αν δεν γίνει κάτι τέτοιο τότε θα έχουμε πολύ αρνητικές επιπτώσεις σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Ευχαριστώ. Στα στοιχεία του Οκτωβρίου αναφέρεται η πίστοση για τα νοικοκυριά. Πέφτει στο μη χρηματοπιστωτικό τομέα. Και συγχρόνως βλέπουμε ε, μεταρρυθμίσεις, διορθωτικές μεταρρυθμίσεις. Εσείς λέτε ότι είναι αναγκαίες, αλλά από ό,τι φαίνεται η συμφωνία για τη χρηματοδότηση του ενιαίου ε, μηχανισμού εξυγίανσης θα είναι για το 2016. Είναι λογικό δεδομένων, τη της κατάστασης κρίσης που ζούμε. Αλλά δεν θα έπρεπε να επιταχυνθεί περισσότερο η κατάσταση. Δεύτερον, λέτε ότι το Fed θα βγει από την διαδικασία μη συμβατικών μέτρων υπολογίζετε τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στην ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική και υπάρχει κάποιος διάλογος, κάποιος συντονισμός. Ο κύριος Δράγκη, με τις επιπτώσεις το, της αγοράς από το ΦΕΔ των κρατικών ομολόγων. Αυτό δεν είναι εύκολα να το διαπιστώσουμε. Έχουμε όμως ένα παράδειγμα, μια εμπειρία που μπορούμε να κοιτάξουμε. Τον Μάιο, αν δεν με πατάει μνήμη μου, φαινόταν ότι το tapering θα μπορούσε να ξεκινήσει ανα πάσα στιγμή, πολύ γρήγορα. Και μαζική μεταφορά ομολόγων στις αγορές. Η κίνηση αυτή είχε να κάνει κυρίως με αναδυόμενες αγορές και πολύ λίγο με την ευρωπαϊκή αγορά ή και τη λεγόμενη non-core αγορά ομολόγων, μη κεντρική. Στις αναδυόμενες αγορές λοιπόν φαίνεται ότι η μετακίνηση αυτή έχει να κάνει με 3, 4, 5 χώρες που ήταν πιο ευάλωτες. Η υψηλό έλλειμμα δηλαδή, ε, χρέος, έλλειψη διευθυντικών μεταρρυθμίσεων κλπ. Αν λοιπόν αυτό το παράδειγμα μπορεί να είναι χρήσιμο, αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να περιμένουμε μεγάλες επιπτώσεις στις δικές μας αγορές ομολόγων, ούτε καν στις λεγόμενες non-core. Από το γεγονός ότι θα σταματήσει η αγορά αυτή ομολόγων. Βέβαια, σήμερα υπάρχει μια βεβαιότητα στις οικονομικές αγορές που είναι μικρότερη από αυτή που είχαμε πριν από μερικούς μήνες. Παρόλα αυτά είναι πολύ δύσκολο να κάνει κανεί προφητείες σε τέτοιου τομεί. Όσον αφορά τώρα το τι μπορούμε να κάνουμε, ρωτάτε αν συνεργαζόμαστε. Στόχος μας είναι η σταθερότητα των τιμών. Θα σταθμίσουμε λοιπόν τη δράση μας ανάλογα με τις επιπτώσεις που θα έχουν όλα αυτά ή ενδεχομένω θα έχουν στην σταθερότητα επί των τιμών. Ευχαριστώ. Και το θέμα της ταχύτητας με την οποία προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις στην Ευρωζώνη και την χρηματοδότηση του ενίου μηχανισμού που είναι για το 26. Τι λέτε, δεν σας φαίνεται πολύ αργός ο ρυθμός αυτός πώς θα ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των αγορών. Τράγκη. Σίγουρα, εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι ο χρόνος που χρειάζεται, και συγγνώμη που δεν σας απάντησα πριν. Λοιπόν, το ένα θέμα είναι το πόσο χρόνος χρειάζεται προκειμένου το ταμείο αυτό να φτάσει στο τελικό 1%. Το άλλο θέμα είναι πότε το Ταμείο, ακόμα και αν δεν έχει ολοκληρωθεί, θα αρχίσει να λειτουργεί σαν ένα πραγματικό Ευρωπαϊκό Ταμείο. Μπορεί κανείς να ξεκινήσει από το βραχυπρόθεσμο. Το να ζητήσουμε από το τραπεζικό σύστημα σε τρία χρόνια να πληρώσει το λογαριασμό είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ γιατί δεν ξέρω ποιες θα ήταν οι συνέπειες. Τον έχουμε όμως ένα ταμείο ακόμα και αν δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν μπορεί να λειτουργήσει πλήρως σαν Ευρωπαϊκό Ταμείο, δεν μπορεί γιατί το πολιτικό μήνυμα θα είναι ουσιαστικό που θα σταλεί. Ευχαριστώ. Ο Γιαπορτφέο από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ να εκφράσω την ικανοποίησή μου. Το 2013 είναι το έτος της εξόδου από το πρόγραμμα προσαρμογής δημοσιονομικό πρόγραμμα που είναι η Ιρλανδία. Το 2014 πιστεύετε ότι θα υπάρξει άλλο κράτος, π.χ. η Πορτογαλία που θα εξέλθει από το πρόγραμμα προσαρμογής. Τι λέτε. Δεύτερο, θα ήθελα να μου πείτε στην περίπτωση του προγράμματος ε, προσαρμογών για μια μεταβατική περίοδο που μπορεί να χρειαστεί για την προσαρμογή στις αγορές. Υπό ποιους όρους ε, και προϋποθέσεις θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι θα, μπορούσε να μπορούσαν να επιβληθούν τέτοιοι όροι και προϋποθέσεις. Μία άλλη ερώτηση σε σχέση με την Τραπεζική Ένωση, σε σχέση με την εποπτεία. Πώς έχει προσεγγίσει το θέμα. Το δεύτερο ερώτημα αφορά με την, την περίπτωση των κρατών που μπορεί να χρειαστούν μια μεταβατική περίοδο ακριβώς ε, για να εξέλθουν από το πρόγραμμα αυτό και να μπορέσουν να βγουν στις αγορές. Υπό ποιου όρους και προϋποθέσεις θα μπορούσαν στο μέλλον να γίνει κάτι τέτοιο και ποιοι όροι και προϋποθέσεις θα επιβαλώνουν για να γίνει κάτι τέτοιο. Το τρίτο ερώτημα αφορά την Τραπεζική Ένωση πώς έχει σχεδιαστεί για την εποπτεία, για την επίλυση προβλημάτων και την διασφάλιση των ε, ε, καταθέσεων η ε, εγγύηση καταθέσεων δεν θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο για μια λύση που θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους πολίτες μας. Και ολοκληρώνω πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε ένα ολόκληρο χρόνο ε, μιας ε, τέτοιας διαδικασίας. Ε, θα ήθελα να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές και το 2014 να μπορούσαμε να δούμε την έξοδο από το πρόγραμμα το δημοσιονομικό ενός ακόμα κράτους της Πορτογαλίας. Ευχαριστώ. Well, thank you. Thank you. Let me say a few words about... Ευχαριστώ. Δύο λόγια για την Πορτογαλία τώρα το, η δέκατη αναθεώρηση του προγράμματος συνεχίζεται. Είναι πολύ πρόημο να πούμε κάτι για τη σημερινή κατάσταση εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων. Πάντως, μέχρι σήμερα η κατάσταση φαίνεται να είναι πολύ κατανοπιτική και οι αρχές δείχνουν να έχουν δεσμευτεί πλήρως την επίτευξη των στόχων. Τα στοιχεία που έχουμε, οι διάφορες δημοσιονομικές μεταβλητές, δείχνουν ότι η κατάσταση βελτιώνεται. Δύο συνεχή τρίμηνα έχουμε αύξηση του ΑΕΠ, η ανεργία πέφτει, έχουμε επίσης καλή απόδοση και των επιτεκείων. Επίσης αυξάνει και επανέρχεται η εμπιστοσύνη. Διαπιστώνεται βελτίωση και στην απόδοση των κρατικών ομολόγων. Βέβαια όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να στηριχθεί και με τη συμμόρφωση στην ερεσιμότητα του προγράμματος. Όσον αφορά τώρα την εφαρμογή κάποιων ε, μέτρων ε, δημοσιονομικής ε, σταθεροποίησης, εδώ διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια μείωση όσον αφορά την απόδοση εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης. Συνεπώς, ενώ η οικονομική κατάσταση βελτιώνεται, μπορεί να χρειαστεί ακόμα χρόνος ώστε να αποδώσει πραγματικά και στον τραπεζικό τομέα. Συνεπώς, ο έλεγχος, η εποπτεία παραμένει ζωτική σημασίας. Και όπως είπα και πριν, είναι πολύ νωρίς να κάνουμε τώρα προβλέψεις για το πότε η Πορτογαλία θα μπορέσει να βγει από το πρόγραμμα. Ιδίω που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η δέκατη αυτή αναθεώρηση. Όσον αφορά την μεταβατική περίοδο, θα υπάρξει πρόγραμμα προσαρμοσμένο στην κατάσταση για το χρονικό αυτό διάστημα και θα δούμε τι μορφή θα πρέπει να πάρει το πρόγραμμα αυτό. Με ρωτήσατε επίσης για την εγγύηση καταθέσεων. Αναβάλλεται με την έννοια ότι θα το συζητήσουμε. Δεν έχει εγκαταληφθεί, αλλά όπως καταλαβαίνετε θα λάβει χώρα κάποια στιγμή στο μέλλον. Τώρα και εγώ σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για τα Χριστούγεννα και συγχρόνως σε όλους σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για τις γιορτές που έρχονται. Πρόεδρος Λέων, εκ μέρους των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ, Σάρον. Δύο ερωτήσεις. Τραπεζική Ένωση και Μακροοικονομία. Πρώτα απ' όλα, Συγχαρητήρια και από μένα όπως και από άλλους για την θέση που υιοθετήσατε όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση, γιατί έτσι μπορούμε να έχουμε μια περίπου ολοκληρωμένη αγορά. Όπως είπατε, έχουμε έναν ενίο μηχανισμό εξυγίανσης και σήμερα κάνατε δηλώσεις υπέρ του μηχανισμού αυτού. Σημαντικό. Όμως για να ολοκληρωθεί η Ένωση αυτή χρειάζεται μια πραγματική Τραπεζική Ένωση. Με τη Σάρων Πήγαμε στο Ενωμένο Βασίλειο με την προσωπία της Επιτροπής μας και είδαμε ότι το ίδιο το Ενωμένο Βασίλειο περιμένει η Ένωση να πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε θέλω να ακούσω ποια είναι η δικιά σας η θέση για τη, τόσα είπε ο κύριος Λικάνεν και για τόσα στηρίξαμε την έκθεση Μακάρθιν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως θα ήταν καλό να υπάρχει μια πραγματική τραπεζική ένωση ώστε να ενοποιούνται όλες οι διαδικασίες. Τώρα, μακροοικονομικά. Ο φίλος Λάγκελ σας ε, είπε, σας ρώτησε, είναι πραγματικά δικιά σας δουλειά να ασχολείστε με τη διαφορετική πολιτική των χωρών μελών. Εντάξει, μια που όντως την Κυριακή δώσατε συνέντευξη, διάβασα τι είπατε και τα παίρνω κατά λέξη. Και λέω κι εγώ ότι είσαστε αυστηρό με τη Γαλλία, όπω και ο συνάδελφο Κλίνη που δεν είναι εδώ μεν τώρα. Και γιατί σα βρίσκω αυστηρό, Γιατί η Γαλλία σήμερα εφαρμόζει μια πολιτική προσφοράς. Είναι έτοιμη να μειώσει το φόρο για τις επιχειρήσεις, μειώνει το χρέος πολύ περισσότερο από την προηγούμενη κυβέρνηση και χρησιμοποιεί και την ευελιξία και ασφάλεια για την αγορά εργασία. Γίνονται λοιπόν διαρθρωτικέ αλλαγέ. Το πραγματικό ζήτημα δεν είναι οι αλλαγές. αλλαγέ. Το είπατε κι εσεί, είναι η δεύτερη ανακοίνωση που κάνατε σήμερα. Είναι ότι υπάρχει απειλή για αποπληθωρισμό. Δεδομένης αυτής της κατάστασης λοιπόν εσεί υιοθετήσατε τα σωστά νομισματικά μέτρα. Αρκούν όμω, γνωρίζετε πολύ καλά την οικονομική ιστορία και η κατάσταση μου θυμίζει λίγο τη συζήτηση που γινόταν τη δεκαετία του 30 στην Επιτροπή Μακμήλαν που γνωρίζετε. Υπήρχε μια γραμμή τότε του Βρετανικού Υπουργείου που έλεγε ότι φτάνει νομισματική πολιτική. Ναι, αλλά τότε δεν υπήρχαν συλλογικέ διαπραγματεύσει, δεν υπήρχε συμβάσει, δεν υπήρχε ελάχιστο μισθό, κοινωνικά μέτρα κτλ. Οπότε η συζήτηση ήταν φτάνει η νομισματική πολιτική ή μήπω πρέπει να προσθεθεί και λίγο δημοσιονομική πολιτική. Αυτό λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω και εγώ τώρα. Δεν υπάρχει εδώ κάποια αντίφαση. Μπορεί να υπάρχει πολυπλησιαστικό φαινόμενο για τα δημοσιονομικά των χωρών και συζητιέται ανάμεσα στο Διεθνές Ταμείο, την Κομισιόν και την ΕΚΤΕ, αλλά δεν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα σε αυτό και το να μιλάμε για μείωση των ε, δαπανών ε, των χωρών προκειμένου να υπάρξει δημοσιονομική εξυγένση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δράγη για την Τραπεζική Ένωση. Υποστηρίζουμε την Τραπεζική Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πάντα βρισκόταν ως υποστηρικτής προς αυτή την κατεύθυνση. Για την έκθεση Λίκανεν είχαμε μια δημόσια διαβούλευση το Μάιο 2013. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από αυτή τη δημόσια διαβούλευση θα κάνει μια μελέτη επιπτώσεων με νομοθετικές προτάσεις που θα αφορούν και το 2013 με εστίαση για την υποχρεωτική διαφοροποίηση των θεμάτων στην έκθεση Λίκανεν και έτσι με την ε, συνεισφορά αυτή στο 2013 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βλέπει ότι είναι επικερδής η διαφοροποίηση διαφορετικών θεμάτων μεταξύ τους και να δούμε εδώ και τον διαχωρισμό των, ε, ε, της χορήγησης υπηρεσιών στους πελάτες. Όμως η συγκεκριμενοποίηση δραστηριοτήτων για τις τράπεζες χρειάζεται σαφώς. Θα πρέπει να υπάρξουν κριτήρια για την υποχρεωτική διαφοροποίηση και τον υποχρεωτικό διαχωρισμό ώστε να υπάρχει μια συνεπής αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι τόσο σημαντικότερο, μια και κάποια κράτη-μέλη ήδη ε, κινούνται ήδη προς ε, την κατεύθυνση διαθωτικών μεταρρυθμίσεων προς αυτή την κατεύθυνση. Καλωσορίζουμε σίγουρα την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προσαρμόσει νομοθετικές προτάσεις για τις διαθωτικές ε, διαφοροποιήσεις και αυτό θα γίνει από ό,τι γνωρίζουμε κατά τα τέλη αυτού του έτους, ώστε να διασφαλιστεί ένα εναρμονισμένο πλαίσιο δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης καλωσορίζουμε τις συστάσεις από την υψηλή ομάδα αξιωματούχων υπό τον Έρκη Λίκανεν ως προεδρεύοντα. Και έτσι καλωσορίζουμε μεν, αλλά θα πρέπει να υπάρχει συνεπές πλαίσιο, ένα ενιαίο συνεπές ε, ε, πλαίσιο, εναρμονισμένο πλαίσιο για, το για τη διαφοροποίηση αυτών των θεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο που είπατε είναι απόλυτα σωστό. Η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να κάνει τα πάντα. Δεν μπορεί να υποκαταστήσει κυβερνήσεις για την απουσία μεταρρυθμίσεων. Δεν μπορεί να ρυθμίσει τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Δεν μπορεί να ρυθμίσει τα προβλήματα τραπεζών που δεν έχουν κεφάλαια Όλα αυτά δεν μπορεί να τα πράξει η νομισματική πολιτική. Η νομισματική πολιτική, η δική μας νομισματική πολιτική συνεισέφερε τα μάλα και έπραξε, έκανε πάμπολα. Και είμαστε έτοιμοι και ικανοί να δράσουμε, αλλά δεν μπορούμε να επιλύσουμε τα πάντα. Δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα άλλων θεσμικών οργάνων. Πρέπει να υπάρξει συνέργεια και αμφίδρομη δράση. Τώρα, για συγκεκριμένα θέματα όσον αφορά την εξυγίανση, η δημοσιονομική εξυγίανση και προπολογισμών. Τώρα, δεν θα πρέπει εδώ να υπονομευθεί η πρόοδος. Και αυτό σαφώς και καλώς εκφράζεται από τις μακροοικονομικές μας προβλέψεις και τα προγνωστικά μας όπου απορρέει σαφώς ότι ένα από τα στοιχεία αυτής της σταδιακής ε, ανάκαμψης θα είναι λιγότερη φορολογική πίεση σε σχέση με τα όσα ίσχυσαν τα, τους προηγούμενους 12 ή 15 ε, μήνες. Αλλά να μην υπονομεύσουμε, να μην οπισθοχωρήσουμε, να έχουμε υψηλότερα χρέη σε υψηλότερα επίπεδα διότι οι αγορές σίγουρα θα δράσουν και θα αντιδράσουν όπως και προηγούμενα αναφέρθηκε σε σχέση με το παράδειγμα που δόθηκε για την Πορτογαλία. Σας ευχαριστώ. Ε, e Ο Γκέι Μίτσελ για το ΕΛΚ από μια ελεύθερη πλέον χώρα. Ναι, ναι, χρειάστηκε πάρα πολύς χρόνος για να αποδεσμευτούμε από τα δεσμά μας, αλλά μην μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες τώρα. Σας ευχαριστούμε κύριε Ντάρκη. Ε, Ντάρκη ε, Δράγη, με συγχωρείτε για την ε, εργασία που έχετε επιτελέσει. Καλά Χριστούγεννα, σε εύχομαι και εγώ. Θα μπορούσατε να μιλήσετε για την Ιρλανδία. Ξέρετε ότι στοικά καταβάλαμε πάρα πολλές προσπάθειες χωρίς να υπάρχει καμία κοινωνική αναστάτωση και εξέγερση. Ουσιαστικά υπομείναμε το ότι μειώθηκαν οι συντάξεις, ότι αυξήθηκαν οι φόροι, το ότι είχαμε υψηλούς φόρους όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, το ότι πολλές φορές χρειάστηκε 10.000 ευρώ κάθε πολίτη ουσιαστικά να δώσει ακόμα και τα παιδιά για την ανεκεφαλοποίηση των τραπεζών και ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε βέβαια το έργο μας αφού το αναγνωρίζω. Βέβαια, ξέρετε ότι καταφέραμε να έχουμε κάποιες επενδύσεις, μειώνεται η ανεργία, καταφέρνουμε επίσης να μειώσουμε το κρατικό μας δημοσιονομικό έλλειμμα και υπάρχουν κάποιες θετικές προοπτικές. Θα πρέπει όμως ο κόσμος πλέον να καταλάβει ότι πραγματικά άξιζαν όλες αυτές οι θυσίες. Το πνεύμα λοιπόν των Χριστουγέννων θα ήθελα να σκεφτείτε λίγο και τους πολίτες της Ιρλανδίας. Πώς θα είναι για αυτούς το 2015 και όλα τα επόμενα έτη ποιο θα είναι ακριβώς, αν θέλετε, το, το τίμημα όλων αυτών των ε, προσπαθειών και των θυσιών. Τι προβλέπετε εσείς για την Ιρλανδία και για όλες αυτές οι υπόλοιπες χώρες, οι οποίες πρέπει να προχωρήσουν σε περαιτέρω δημοσιονομική εξυγίανση τόσο κατά το 2014 όσο και τα επόμενα έτη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, Εξετάζοντας την Ιρλανδία έχετε απόλυτα δίκιο. Η εφαρμογή του προγράμματος στην Ιρλανδία ήταν και παραμένει ε, πάρα πολύ καλή, ακολουθεί δηλαδή το αρχικό πρόγραμμα, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε το φυστάμενο πρόγραμμα με ιδιαίτερη επιτυχία. Ωστόσο, όταν ατενίσουμε το μέλλον, βλέπουμε ότι ε, υπάρχει μια θετική, αλλά πιο προσεκτική, αν θέλετε, συντηρητική αποτίμηση του προπολογισμού για το 2014, μολονότι θα επιτευχθούν κάποιοι στόχοι. Τώρα, όσον αφορά τον λόγο ελλείμματος προς το ΑΕΠΑ, 4,8% προβλέπεται ότι θα είναι, όπου ουσιαστικά έχουμε καλύτερη, καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη που είχε γίνει για 5,1%. Ο τραπεζικός όμως κλάδος της Ιρλανδίας δημιουργεί ακόμα κάποιες ανησυχίες. Υπάρχουν κάποια κρεμή προβλήματα τα οποία θα πρέπει πολύ γρήγορα να επιληθούν. Πρόσφατα είχαμε κάποια αποτελέσματα όσον αφορά την αξιολόγηση των ισολογισμών των τραπεζών της Ιρλανδίας και είδαμε ότι δεν υπάρχει κεφαλιακή ανεπάρκεια μεν, αλλά θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές όσον αφορά τις ε, προμήθειες για συγκεκριμένα στοιχεία του ενεργητικού και θα πρέπει να καλυφθούν οι ανεπάρκειες αυτές προτού γίνει συνολική αξιολόγηση από τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό. Πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι η αξιολόγηση που έχει γίνει από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή δεν είναι οριστική και ότι θα πρέπει να προσβλέπουμε προς μια ολοκληρωμένη επιτυχία αξιολόγηση από τον ενιαίο αποπτικό μηχανισμό. Η έξοδος λοιπόν της Ιρλανδίας από το πρόγραμμά της καταδεικνύει τελικά το ότι έπρεπε να αναλυφθούν κάποια μέτρα, ότι έπρεπε να υιοθετηθούν κάποιες συγκεκριμένε δράσεις. Και αυτό για τους εξής λόγους. Ε, ποιο θα είναι το αντίκρισμα για τον ε, πληθυσμό. Κοιτάξτε, μεγαλύτερη ανάπτυξη, περισσότερες θέσεις απασχόλησης και περισσότερη ελευθερία, αν θέλετε. Νομίζω ότι κάποιος στην Ιρλανδία σήμερα έκανε μια δήλωση και είπε ότι ανάκτησε την εθνική της περηφάνεια η χώρα βγαίνοντα από το πρόγραμμα. Αληθεύει αυτό, σωστή η δήλωση, αλλά αυτό ουσιαστικά στην πράξη ισχύει αν όντω μεταφράζεται σε υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη και περισσότερε θέσει εργασία. Σα ευχαριστώ. Ο Πίτερ Σκίνερ, σοσιαλιστέ. Ουσιαστικά λέτε ότι είμαστε στην αρχή μιας ε, επιτυχίας με όλα όσα πέρασαν οι Ιρλανδοί, τους αξίζει ότι καλύτερο. Άκουσα και τα σχόλιά σας κύριε Τράγκη για την αξιολόγηση ομολόγων ε, ενεργητικού και γενικά το νέο ρόλο της ΕΚΤ. Όμως εξακολουθείτε να είσαστε Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οπότε ο έλεγχος που κάνετε και φιλοσοφικά οι προθέσεις σας ποιες είναι ακριβώς. Δεν μπορεί να ασχοληθείτε με τα μακροοικονομικά αν δεν ασχοληθείτε και με την εποπτή επιτόπου. Έχετε τρεις εποπτικές αρχές οι οποίες μέσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου παίζουν το ρόλο τους Δεν θέλω να πω ότι δεν έχει γίνει προσπάθεια, αλλά αν βλέπω τα αποτελέσματα, είμαστε μόνο στην αρχή και ό,τι συνταγές βρήκαμε νωρίτερα έχουν ξεπεραστεί από τα γεγονότα. Δεν ξέρω, συνεπώς, ποιο ρόλο πιστεύετε ότι θα πρέπει να παίξουν τα εποπτικά μέσα και τα μακροοικονομικά που διαθέτουμε. Πώς θα υπάρξει διαφοροποίηση, πώς θα ακούσετε τους μεν και τους δε, πώς θα διασφαλίσουμε ότι λαμβάνετε υπόψη το τι πρέπει να γίνει κάθε φορά, που θα πούν οι υποπτικοί μηχανισμοί, οι μακροοικονομικοί, το τι πρέπει να γίνει. Τράγκη. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση και την αντιμετωπίσαμε από βράση του Συμβουλίου μας. Ε και παρότι δεν έχει αναγγελθεί ακόμα έχει προσεγγιστεί με τρόπο ώστε οι δυνατότητες εποπτείας θα οδηγήσουν στο να συγκεραστούν με τις ε, μακροοικονομικές ε, ευθύνες μας. Δεν είναι εύκολο αυτό το θέμα να επιληθεί. Θέλουμε να έχουμε ε, διαφοροποίηση μεταξύ εποπτείας και νομισματικής πολιτικής. Από την άλλη πλευρά όμως για την εποπτεία κονδυλίων υπάρχουν συνέργειες που και αμφότερες οι πλευρές μπορούν να κερδίσουν από αυτή τη δραστηριότητα εντοπισμό και ανείχνευση προβλημάτων, εντοπισμός ε, φούσκας ε, σε συγκεκριμένα πεδία. Με ποια πολιτική θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα τέτοιο πρόβλημα και πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Υπάρχει λοιπόν μια εξειδικευμένη προσέγγιση και αντιμετώπιση από το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό και ταυτοποίηση των επιμέρους ε, και πριν από τα τέλη του έτους θα, μπορέσουμε να τα γνωστοποιήσουμε. Η ιδέα όμως είναι ακριβώς αυτή η οποία προτείνατε εσείς, δηλαδή να μπορέσουμε να ασκήσουμε μακροπρόθεσμα την εποπτεία με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε εποπτεία μακροπρόθεσμης διάρκειας ώστε να έχουμε ανταλλαγή πληροφοριών να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες ώστε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τη σοβαρότητα καταστάσεων. Ευχαριστώ. Δεν είναι εδώ ο Φαμπρίτσιο. Άστριτ Λούλιν. Ευχαριστώ. Κύρια Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε Τράγκη, Ξαναβλέπουμε το ευρωπαϊκό εποπτικό σύστημα. Τα αναθεωρούμε. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν κάποιοι συνάδελφοι επαναλαμβάνουν την επιθυμία. Η ΕΚΤ, μάλλον διαπιστώνουν ότι η ΕΚΤ συσσωρεύει υπερβολικά πολλές εξουσίες. Γιατί υπάρχει νομισματική πολιτική, υποπτική μηχανισμοί και βρίσκουν ότι όλα αυτά είναι πολλά για ένα μόνο θεσμικό όργανο. Διότι οι ρήτρε ασφαλείας, από ό,τι φαίνεται, δεν τους πείθουν ότι φτάνουν. Εσείς λοιπόν, Πρόεδρε, τι επιχείρημα έχετε για να τους απαντήσετε. Πιστεύετε ότι τελικά οι ανησυχίες τους θα αποδειχθούν βάσιμες ή ότι υπάρχει μια κατάλληλη διακυβέρνηση ώστε να αντισταθμίσει τις φιλοδοξίες και τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πρόεδρος Δράγκη, ευχαριστώ. Να πω πρώτα απ' όλα ότι δεν είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που ζητάει τη συσσόρευση αυτών των εξουσιών. Εσείς οι νομοθέτες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή και το Συμβούλιο το ζητάτε. Εσείς αποφασίσατε ότι ο καλύτερος ε, φυσικός χώρος για τον ενίο εποπτικό μηχανισμό ήταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εγώ τι έχω να απαντήσω. Ότι απαντάω πάντα. Ότι δηλαδή θέλουμε η λογοδοσία να είναι όσο γίνεται ε, περισσότερη, να υπάρχει διαφάνεια για να υπάρχει έλεγχος. Εμείς έχουμε συμπεριλάβει τόσο ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι δηλαδή ο καλύτερος τρόπος είναι να δεχτούμε υψηλότερες προδιαγραφές λογοδοσίας από ό,τι έχουμε για την νομισματική πολιτική μέχρι τώρα. Και αυτός είναι και ο στόχος της διοργανικής συμφωνίας. Ότι δηλαδή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι αυτό ένα πολύ σημαντικό βήμα για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γενικά και ειδικότερα την Οικονομική Επιτροπή και την Πρόεδρό τη. Ευχαριστώ πολύ Σάρων, για όλα όσα και εσύ και οι συνεργάτε κάνανε για να επιτευχθεί αυτή η διοργανική συμφωνία. Εκτός μικροφώνου παρέμβαση της κυρίας Λούλινγκ. Πρόεδρος, Ρεμόν Τρεμόζα εκ μέρους της Άλντε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ντράγκη, μια πολύ, κάποιες πολύ σύντομες ερωτήσεις. Νομίζετε ότι είναι σύμβατα όλα αυτά με την Τραπεζική Ένωση, με τη δυνατότητα των κρατών μελών να συνεχίσουν να έχουν δικαίωμα αρνησή ε, κατά των ευρωπαϊκών αποφάσεων για να, πώς είπατε κύριε, να εξακολουθούν να έχουν το δικαίωμα αρνησή το βέτο που θα μπορούν να, να ασκήσουν. Συγγνώμη για τα άσχημα αγγλικά μου στην προφορά μου, λέει ο μιλητής. Και μετά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μια σφαιρική αξιολόγηση, αντιμετωπίζουμε αβεβαιότητα και ανασφάλεια. Αυτό είναι κύρια ανησυχία, επειδή σημαντικές παράμετροι δεν έχουν ακόμα ακόμα γνωστοποιηθεί. Για παράδειγμα σε σχέση με το κρατικό χρέο, το εύρο των δοκιμασιών τραπεζών, ε, τι θα γίνει με το συστημικό ε, κίνδυνο και ποιο είναι αυτό. Ε. Και μέσα στα λίγα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μα, φυσικά δεν μπορούν όλα αυτά να αποσαφινιστούν. Αλλά τουλάχιστον πείτε μα ποια χρονική στιγμή θα γνωρίζουμε και θα μάθουμε ποια θα είναι η αντιμετώπιση του κρατικού χρέους ε, και το εύρος ε, των ε, τραπεζικών δοκιμασιών από πλευράς τεστ. Σε ποιο δικαίωμα αρνησή κυρίας αναφερθήκατε κύριε, των κρατών μελών λέει ο μιλητής, που φαίνεται ότι στη νέα συμφωνία για την επίλυση προβλημάτων οι κυβερνήσεις των κρατών μελών θέλουν να συνεχίσουν να έχουν δικαίωμα αρνησή κυρίας κατά μιας ευρωπαϊκής απόφασης που θα λαμβάνεται για την επίλυση τραπεζικών θεμάτων. Δεν γνωρίζω κάτι παρόμοιο, λέει ο κύριος Δράγκη. Μπορεί να συμβαίνει ίσως αυτό, αλλά δεν έχω συνειδητοποιήσει να, ότι αυτό είναι πράγματι αυτό το οποίο υφίσταται. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει, δεν το γνωρίζω. Αλλά αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, τι θα λέγατε αν κάποια κράτη-μέλη θα είχαν μια τέτοια ικανότητα άσκησης άρνηση όχι, δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν. Δεν νομίζω ότι θα είχε νόημα μάλιστα κιόλα να έχουν δικαίωμα άρνηση όταν θα δηλώνεται μια τράπεζα θα πιστοποιείται ως μη βιώσιμη και να ασκούν δικαίωμα άρνηση από πλευρά τους. Το θέμα της άρνηση μπορεί να αναφύεται τότε και αν όταν ε, οι ε, πόροι και οι ικανότητες του ESM θα ε, χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος, για την επίλυση ενός προβλήματος με δράσεις. Σε αυτή την κατάσταση έχουμε την υφιστάμενη συνθήκη του ESM, τη συμφωνία, που κάθε ένας από τους εμπλεκόμενους έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας. Αλλά για την συνολική αξιολόγηση μη βιωσιμότητας μιας τράπεζας δεν έχω υπόψη μου να υπάρχει δικαίωμα αρνησικυρίας από κάποιους. Το δεύτερο σημείο που αναφέρατε, από ό,τι γνωρίζω, σίγουρα έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει ένα βαθμό αβεβαιότητα και ανασφάλεια. Αλλά μόλι ξεκινήσαμε, είμαστε στα σπάργανα, στα πρώτα βήματα. Πρέπει να επιταχύνουμε την ε, αποσαφήνιση των παραμέτρων αυτών ε, όσον αφορά τα τεστ, ε, τη δοκιμασία που θα υποστούν οι τράπεζε. Και όσο καλύτερα και πιο γοργά γίνουν αυτά, τόσο καλύτερο θα είναι το αποτέλεσμα. Τώρα να μην ξεχνάμε βέβαια και κάτι άλλο στη συνέχεια ότι παρότι το τελικά, τα τελικά αποτελέσματα αυτών των δοκιμασιών θα αναγγελθούν το Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο του χρόνου 2014 αν στο μεσοδιάστημα εντωμεταξύ θα είχαμε κάποια δράση που θα αναλαμβανόταν είτε να ανακεφαλαιοποιηθούν ή να αποκτήσουν κεφάλαια κάποιες τράπεζες επειδή θα είχα, είχε διαπιστωθεί ότι απουσίαζαν ή υπήρχε απουσία τέτοιων, τέτοιας επαρκούς κεφαλαιοδότησης αυτό ισχύει για, δι, για, για κάποιες δημόσιες κρατικές εταιρείες θα ήταν κάτι απίθανο να αναμένουν μέχρι τον Οκτώβριο 2014 προτού γνωστοποιηθούν όλα αυτά για να μπορέσουν να δράσουν πιο πριν. Αν λοιπόν διορθωτική δράση θα έπρεπε να αναλυφθεί, ιδιαίτερα σε σχέση με κρατικές εταιρείες, αυτά θα έπρεπε άμεσα να γνωστοποιηθούν και να τα γνωρίζουν, διότι οι αγορές θα πρέπει να γνωρίζουν όλες αυτές τις παραμέτρους και στοιχεία. Θα επιταχύνουμε λοιπόν την επικοινωνία και επ' αυτών των στοιχείων το δυνατόν όσο, όσο γίνεται περισσότερο. Τα τελικά αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν τον Οκτώβριο του 2014. Εντάξει, αλλά αληθεύει επίσης ότι για διάφορες περιπτώσεις και ανάλογα με το ότι διαπιστώσουμε οι κανόνες και οι κανονισμοί της αγοράς θα απαιτήσουν άμεση ενημέρωση και πληροφόρηση αν διορθωτική δράση θα πρέπει να αναλυφθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Μπαλντίνη εκ μέρους των Σοσιαλιστών. Κύριε Πρόεδρε, θα θέσω ένα πρώτο ερώτημα ως νέος Ευρωβουλευτής από την 1η Ιουλίου, από την Κροατία προέρχομαι, ξέρετε ότι πολλές φορές ενώ συζητάμε με ευρωσκεπτικιστές, ιδίως κατά το δεύτερο τμήμα του τρέχοντος έτους, είδαμε κάποια παραδείγματα της θετικής δράσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πομένως σας συγχαίρω για τα θετικά αυτά αποτελέσματα, για τη θετική σας δράση. Θα ήθελα παρόλα αυτά να θέσω ένα ερώτημα, βασιζόμενος κυρίως ε, στο... στη θετική έκβαση του προγράμματος της ε, Ιρλανδίας. Ενδεχομένως να είναι πολύ πιο εύκολο να βγει κανείς από αυτό το καθεστώς οικονομικής κρίσης στις πιο μικρές τελικά χώρες, στις χώρες εκείνες που έχουν πιο μικρή οικονομία, όχι τόσο σημαντική όπως κάποιες άλλες ε, χώρες, όπως για παράδειγμα της Νότιας Ευρώπης. Όσον αφορά την ε, περιοχή τη δική μου, πρέπει να σας πω ότι εμείς ε, βλέπουμε ότι έξι συγκεκριμένες περιοχές στην χώρα μου είχαν μια σημαντική Μάλλον έξι χώρες είδαμε ότι πολύ, είχαν πολύ σημαντική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη. Από την άλλη έχουμε χώρες όπως η Κροατία, η, η Σλοβενία, που έχουν πολύ σημαντικά προβλήματα, ιδίως στον τραπεζικό τομέα. Βρισκόμαστε στο τέταρτο κατά, τέταρτο κατά συνέχεια τρίμηνο μείωση της οικονομικής ανάπτυξης στην Κροατία και μολονότι παρουσιάζουμε εμεί μια σημαντική οικονομική ανάπτυξη σε σχέση με την υπόλοιπη περιοχή, έχουμε πολύ σημαντικά προβλήματα οικονομική ανάπτυξη παρόλα αυτά. Θα μπορούσατε να κάνετε κάποιε συστάσει οικονομική φύσεω ή συμφωνείτε κι εσεί με αυτό το οποίο είπα πριν από λίγο, ότι θα έπρεπε οι χώρες αυτές, οι οποίες αναφέρθηκαν, να μπουν και αυτές σε έναν δρόμο οικονομικής ανάπτυξης εξόδου από τις κρίσεις όπως η Ιρλανδία. Κύριος Δράγκη, κοιτάξτε, μπορούμε να έχουμε μία κάποια συγκρατημένη αισιοδοξία σήμερα, ατενίζοντας όντως το παράδειγμα της Ιρλανδίας, όχι μόνο της Ιρλανδίας όμως, αλλά και της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, η οποία είναι μεγαλύτερη χώρα και η χώρα αυτή έχει επιτύχει τεράστια πρόοδο. Όλες αυτές οι χώρες έχουν σημειώσει πολύ σημαντική πρόοδο. Δείτε πώς ήταν η κατάσταση στις χώρες αυτές πριν από ένα-ενάμιση χρόνο. Και δείτε ποιες σημαντικές αλλαγές έχουν γίνει στις χώρες αυτές, θετικές αλλαγές. Η Ελλάδα είναι ένα ακόμα θετικό παράδειγμα. Το γενικότερο λοιπόν αίσθημα είναι ότι ανεξάρτητα από το μέγεθος της χώρας, αν ακολουθούν τις σωστές πολιτικές, τότε μπορεί κανείς να ξεπεράσει την κρίση. Οι χώρες αυτές μπορούν να βγουν από την κρίση μπορούν να υπερβούν, αν θέλετε, αυτό το δύσκολο μεγάλο εμπόδιο που έχουν μπροστά του, στην κρίση, μπορούν να διαβούν το ποτάμι αυτό και μπορούν να αποφεληθούν από όλα αυτά τα ωφέλη, δηλαδή μεγαλύτερη απασχόληση, μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη. Πρέπει όμω να καταδείξουν αποφασιστικότητα όταν προσπαθούν να διορθώσουν τα δύναμα σημεία των οικονομιών του που οδήγησαν σε αυτέ τι ανισορροπίε. Σα ευχαριστώ. Okay, thank you very much. Πρόεδρος, Ευχαριστώ. Δεν έχω άλλους στον κατάλογό μου. Αλλά επειδή έχουμε λίγα λεπτά ακόμα, αν υπάρχει κάποιος άλλος που καίγεται να ρωτήσει κάτι. Ε, ναι, βέβαια. Δεν ξέρω ότι μπορούσα να βασιστώ σε σένα για την τελευταία ερώτηση. Ο κύριο Βέρνερ Λάγκεν, έχω ακόμα μια ερώτηση προ τον κύριο Πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Τα stress tests, οι δοκιμασίε, τα τεστ τραπεζών, το αναφέρατε σε σχέση με την εποπτεία τραπεζών. Ρίχνουν τη σκιά του αυτέ οι δοκιμασίε Μια και δεν είμαστε σε θέση να έχουμε μια αξιολόγηση των κρατικών ομολόγων, τώρα στρέφονται τα βλέμματα όλων για το πώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αντιμετωπίσει αυτό το μεγάλο πρόβλημα τη στάθμισης και αξιολόγηση των κρατικών ομολόγων όσον αφορά τους κρατικούς ισολογισμούς. Και τι θα κάνετε σε σχέση με την επιτυχία εκείνων των αξιολογήσεών σας και των αξιολογήσεων των κυβερνήσεων σε σχέση με μια σειρά προγραμμάτων, την τον διαφοροποίηση του κρατικού χρέους και του τραπεζικού χρέους. Δυστυχώς δεν βλέπω να γίνεται κάτι τέτοιο ακόμα. Yeah. Υπάρχουν δύο διαφορετικά θέματα εδώ. Το ένα είναι η αξιολόγηση των ομολόγων για τον τρόπο που λειτουργήσαν και από την άλλη μεριά είναι να ζυγίσουμε τους κινδύνους των διαφόρων κυβερνητικών ομολόγων. Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει συνολικά να συζητηθούν στην Επιτροπή Βασιλείας. γιατί μπορεί κανείς να πει ότι πρέπει να υπάρχει χωριστός ε, χειρισμός για τα βρετανικά ομόλογα σε σχέση με τα αμερικανικά, τα βρετανικά ή τα κινέζικα ανά τον κόσμο. Γιατί αλλιώς βάζετε τις τράπεζες της Ευρωζώνης σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σύγκριση με τις αμερικανικές, ιαπωνικές ή κινέζικες τράπεζες. Οπότε προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα συζητηθούν τα ομόλογα που πιστεύουμε ότι είναι η Επιτροπή της Βασιλείας. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ε, λαμβάνουμε υπόψη μας και τα, κυβερνητικά, τα κρατικά ομόλογα στα τεστ αντοχής. Όπως οποιοδήποτε άλλο ενεργητικό που ανήκει στις τράπεζες, έτσι εξετάζονται και τα ομόλογα αυτά, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται ε, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Άρα λοιπόν, άλλο είναι ο στάθμιση κινδύνου για τις τράπεζες και για τα κρατικά ομόλογα και άλλο είναι πόσα κρατικά ομόλογα ανήκουν σε τράπεζες οι οποίες βρίσκονται στην Ευρωζώνη και πώς συμπεριφέρονται τα ομόλογα αυτά κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής αντοχής. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Α, ακόμα κάποιος. Κύριε Ντράγκη, το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση, γράφει μια εικόνα όχι και τόσο ενθαρρυντική. έχετε κάτι στο μυαλό σας που μπορείτε να κάνετε ένα νέο MTRO, νούμερο 2 δηλαδή, και τι επιπτώσει θα έχει αυτό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η παρούσα κατάσταση είναι τέτοια όπου οι τράπεζες επιστρέφουν τα LTRO, τα Long Term Refinance Operations. Οπότε, Ας αναρωτηθούμε γιατί δεν δανείζουν οι τράπεζες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τρεις είναι οι λόγοι. Ο ένας είναι ότι δεν έχουν αρκετή χρηματοδότηση, οι ίδιες, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίσαμε πριν από δύο χρόνια με τα LTROs, γι' αυτό και οι τράπεζες επιστρέφουν τα χρήματα. Οπότε πριν φάτσε δεν υπάρχει ε, θέμα έλλειψης χρηματοδότησης, να είναι αυτό δηλαδή το κύριο εμπόδιο, ο λόγος για τον οποίο δεν δανείζουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έπειτα υπήρξαν και οι ασφάλειες ομολόγων. Όπως είπα και πριν, οι καταθέσεις συνολικά στις non-core χώρες έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Άρα δεν είναι έλλειψη χρημάτων. Τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο δεν φαίνεται να είναι το κύριο πρόβλημα. Δεύτερος λόγος. Δεν υπάρχει αρκετό κεφάλαιο. Τώρα εδώ αυτό θα το διαπιστώσουμε με τα τεστ αντοχής. Αλλά μην ξεχνάμε ότι από το 2008 μέχρι σήμερα, από το 2008-2009 μέχρι το τέλος του 2012 αν δεν απατώμε, πάνω από μισό τρισεκατομμύριο ευρώ προσθέθηκε στο κεφάλαιο των τραπεζών. Το μισό ήταν ε, δημόσιο χρήμα και το μισό από τον ιδιωτικό τομέα. Και πολλά χρηματοπιστωτικά ε, ιδρύματα έχουν αυξήσει το κεφάλαιό τους και τους τελευταίους 5-6 μήνες, που είναι καλό, θετικό, πολύ καλή εξέλιξη. Συνεπώς, να και μάλιστα εδώ μιλάμε για τον μεσόρο, έτσι. Εννοείται ότι υπάρχουν χιλιάδες τράπεζες και μπορεί να έχουμε διαφορετική πραγματικότητα στις μεγάλες και στις μικρές τράπεζες. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτός ο μέσος όρος, πάντως είναι ένας μέσος όρος. Έλλειψη κεφαλαίου μπορεί να είναι πρόβλημα για μια κατηγορία τραπεζών, παρόλο που συνολικά δεν το βλέπουμε αυτό σαν πρόβλημα. Ο τρίτος πάντως λόγος είναι ο κίνδυνο, η εξολόγηση κινδύνου. Οι τράπεζε δεν δανείζουν γιατί φοβούνται ότι δεν θα ξεπληρώσουν τα δάνειά τους οι πελάτες τους. Και οι πελάτες δεν ε, ξεπληρώνουν γιατί δεν βρίσκουν που να πουλήσουν το προϊόν τους. Έπειτα, αυτός ήταν ο πρώτος λόγος στην έρευνα που κάναμε, όχι την τελευταία, την πρώτη τελευταία έρευνα που κάναμε στι μικρομεσαίες επιχειρήσει όπου του ρωτήσαμε ποιο είναι το κύριο εμπόδιο για σας να προχωράει η επιχείρησή σας. Και είπαν έλλειψη πελατών. Αυτό ήταν το κύριο. Η έλλειψη κεφαλή ήταν το δεύτερο. Αυτό τώρα θα βελτιωθεί. Θα φανεί αυτό σύντομα. Ότι δηλαδή η έλλειψη εμπιστοσύνη των τραπεζών στους πελάτες θα μειωθεί. Τι μου λέτε, μου κάνετε νόημα, το βλέπω, είσαστε έτοιμοι, ναι, τη βλέπω την πίεση να μου έρχεται από εσά ότι πρέπει να τελειώσω. Πρόεδρος, όχι, η Σιλβή θέλει κάτι να ρωτήσει. Ευχαριστώ Σαρών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μια ερώτηση ακόμα. Αφαντήσατε. με μεγάλη πειθό όσον αφορά την έξοδο από το ευρώ. Εγώ θέλω να σας ε, ζητήσω να αντιδράσετε στην ανησυχία που έχω όσον αφορά την αμοιβή εμπιστοσύνη στην Ευρώπη και για το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στο βορρά και το νότο, παρά τις προσπάθειές σας, παρά την ομοθεσία που έχουμε εγκρίνει, τι μπορούμε να κάνουμε ως θεσμικά όργανα για να μην μεγαλώσει το χάσμα αυτό Νομίζω εγώ ότι αποτελεί μέρος της δικιάς σας εντολής, γιατί πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη. Και αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των διαφόρων φορέων του συστήματος, τότε τα τεχνικά στοιχεία που εσείς ε, ε, προτείνετε δεν θα έχουν το αποτέλεσμα που εμείς περιμένουμε. Νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση που βάζετε, διότι η εμπιστοσύνη πράγματι είναι στην καρδιά του ζητήματος σε επίπεδο διακυβέρνησης στην Ευρώπη. Οπότε, ας αναρωτηθούμε, γιατί εξαφανίστηκε η εμπιστοσύνη. Εξαφανίστηκε γιατί οι άνθρωποι είχαν την αίσθηση είτε ότι οι κανόνες δεν τηρούνται, η δημοσιονομική πειθαρχία, δηλαδή του συμφώνου σταθερότητα ήταν κάτι που είχε ξεχαστεί στην αρχή της δεκαετίας του 2000 ή επειδή ο κόσμος ένιωσε ότι δεν έγιναν διορθωτικές μεταρρυθμίσεις με την εξαίρεση μιας δύο χωρών. Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν να επανέλθει η πιστοσύνη είναι η συμμόρφωση προς τους συμφωνημένους κανόνες και οι οικονομικές πολιτικές εννοείται ότι έχουν επιπτώσεις και στο διπλανό μας. Βλέπετε, έλλειψη εμπιστοσύνη υπάρχει εξαιτία τη αδιαφορία μερικέ φορέ των πολιτικών αποφάσεων που δεν σκέφτονται αυτοί που τις παίρνουν ότι οι αποφάσεις αυτές επηρεάζουν και τους άλλους. Αγνοούν ή τέλο πάντων αμελούν το γεγονός ότι υπάρχουν επιπτώσεις και στις γείτονες χώρες. Συνεπώς οι πολιτικές που υιοθετούνται πρέπει να είναι τέτοιες ώστε οι χώρες να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους από μόνες τους. Δεν μπορεί να προειδοποίηση ότι θα έχουμε μονίμως κάποιους που θα βάζουν χρήματα και κάποιους που θα χρωστάνε χρήματα. Πρέπει να δείξουμε ότι κάποια στιγμή όλες οι χώρες μπορούν να γίνουν ο πιστωτής αυτός που δίνει χρήματα αντί να παίρνει. Έτσι θα επανέλθει η πιστοσυνη Πρόεδρος, ευχαριστώ. Άντε, άλλος ένας η Περβάνς Μπέρες. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Έχετε κάνει πολλά πράγματα, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, υπουργοί οικονομικών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από την αρχή της θητείας κινητοποιήθηκαν προκειμένου να εξασφαλίσουμε την σταθερότητα των αγορών και προκειμένου να αυξηθεί και η εμπιστοσύνη στην οποία αναφερθήκατε. Υπάρχει όμως και το ζήτημα της χρηματοδότησης οικονομίας. Αναφερθήκατε σε αυτό πριν από λίγο, τα μιλήσετε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ιδίω τον κύριο Μπαρνιέ υποβάλλει πλέον ένα κείμενο το οποίο αναφέρεται στο ζήτημα της ε, μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης των επενδύσεων. Βλέπουμε ότι σε χώρες όπως η Γερμανία, Ινστιτούτα όπως το ΔΙΦ θεωρούν ότι 75 ε, δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως απαιτούνται προκειμένου να καταφέρουμε να κάνουμε τις απαραίτητες επενδύσεις, να χρηματοδοτήσουμε τις απαραίτητες επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα γίνει κάτι τέτοιο και πώς μπορείτε εσείς να συμβάλλετε μέσω της νομισματικής πολιτικής γιατί νομίζω ότι ε, έχουν εγκριθεί πολλοί κανονισμοί και πολλές νομοθεσίες που έχουν επίπτωση στον τομέα αυτό. Κοιτάξτε, η σημαντικότερη συμβολή που μπορεί να επιφέρει νομισματική πολιτική είναι να συνεχίσει να επιτελεί το βασικό της έργο, σταθερότητα των τιμών. Και όταν λέω σταθερότητα των τιμών, το είπα και αυτό πριν από λίγο, αναφέρομαι και στις δύο κατευθύνσεις, και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχουμε ένα πληθωρισμό, ο οποίος είναι πολύ χαμηλός, γύρω στο 2% για παραταταμένη χρονική περίοδο. Επομένως, θέλουμε να έχουμε μια νομισματική πολιτική, η οποία θα είναι προσαρμοστική στη ζήτηση. Γι' αυτό λόγο έχουμε κάνει μελλοντικές προπτικές όπου λέμε ότι τα επιτόκια θα είναι για παραταμένο χρονικό διάστημα σε χαμηλά επίπεδα, Αναλάβαμε δράση τον Νοέμβριο σύμφωνα με αυτό το forward guidance, μειώσαμε τα επιτόκια και θα συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ποιοι είναι οι κίνδυνοι που ενυπάρχουν σε αυτόν τον πολύ χαμηλό πληθωρισμό και έχουμε στη διάθεσή μας πολλά μέτρα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αν χρειαστεί. Νομίζω ότι αυτή είναι η σημαντικότερη συμβολή της νομισματικής πολιτικής. Ευχαριστώ. Okay, thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώνεται λοιπόν ο διάλογός μας. Θα είστε σύντομα πάλι μαζί μας, επομένως προσβλέπουμε στην επόμενη ανταλλαγή απόψεων που θα έχουμε. 3η Μαρτίου, μάλιστα. 3 Μαρτίου 2014. Έχουμε ήδη προγραμματίσει λοιπόν την ε, επόμενη μας αυτή συνάντηση. Ο Βέρνερ. Επιτρέψτε μου την παρουσία του Προέδρου να κάνω μια παρατήρηση επί διαδικαστικού για τον κανονισμό την Πέμπτη το πρωί στην Ολομέλεια. Σχεδόν ε, με κενή Ολομέλεια είχαμε την ετήσια έκθεση του 2012 που συζητήσαμε. Το βρήκα κατεσχήνη σε σχέση με το Ευρωκοινοβούλιο. Ε, έσχος αυτό. Και παρακαλώ να αποστείλετε επιστολή στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σούλτς, και να του πείτε ότι όπως και σε άλλες σημαντικές εκδηλώσεις δεν μπορούν ταυτόχρονα να, γίνονται τριμερείς διάλογοι, ε, συναντήσεις προεδρίου κτλ. Παρακαλώ παρακαλώ η Πρόεδρος να δραχθεί της ευκαιρίας και να αποστείλει επιστολή στον Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου σε σχέση με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Uh, ναι. Πράγματι είχα ήδη μια συζήτηση με τον Πρόεδρο Σούλτς και για αυτά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα. Εν μέρει επειδή πολλοί τριμερεί ε, διάλογοι ε, βρίσκονται υπό εξέλιξη, όχι μόνο σε αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή, αλλά και σε άλλε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ. Και είχαμε και αυτό το θέμα το οποίο ε, σε σχέση με την τραπεζική οδηγία και αυτό δημιουργεί μείζον πρόβλημα. Βέρναρ και πάλι. Θέλω να υπενθυμίσω ότι την Τρίτη, την Τρίτη, την Τρίτη είχαμε ένα πρόγραμμα μέχρι τις 11.30 και μετά ξεκινήσαμε με τις ψηφοφορίες ψηφίζοντας με 45, 45 λεπτά πριν από το προβλεπόμενο τέρ, τέλος είχε ολοκληρωθεί η συζήτηση και έκλεισε η Ολομέλεια. Τερματίστηκαν οι εργασίες. Αυτό το σχεδιασμό εργασιών τον θεωρώ λέθριο. Δεν μπορώ να συζητήσουμε εδώ για την Ολομέλεια. Έχουμε άλλα θέματα. Σε επίπεδο συντονιστών θα έπρεπε να τεθεί. Τώρα ο Πάμπλο να λαμβάνει την Προεδρία για την υπόλοιπη σημερινή συνεδρίαση. Και αποχαιρετάμε εδώ τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Continuamos con el orden del día, punto 5 de la agenda. Συνεχίζουμε την ημερήσια διάταξη, σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Παρουσίαση του σχεδίου έκθεση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Εισηγητή για αυτό το θέμα είναι ο κύριος ε, Φιλίπ Ντεμπάκερ. Δίνω αμέσως λοιπόν τον λόγο στον κύριο Ντεμπάκερ, παρακαλώ. Yes, yes, thank you, President. Um... Ευχαριστώ, Πρόεδρε αγαπητοί ευρωβουλευτές δεν θα ξεκινήσω διαβάζοντας όλη την έκθεση η έκθεση αυτή νομίζω είναι και μέρος αυτής της συζήτησης που ήδη την είχαμε αρκετές φορές με τους κοιόδης συζητητές για να δούμε προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούν οι συστάσεις για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής. Και είχαμε και συζητήσεις κατά το παρελθόν σχετικά. Αυτό που θα κάνω είναι σε σχέση με την ε, έκθεση αυτή που είναι σαφέστατη επιτρέπει από το δυνατόν περισσότερες κοινοβουλευτικές ομάδες να εμπλακούν και να συμμετάσχουν. Αυτό που προσπάθησα εγώ να κάνω είναι ευθύ εξ αρχής να διασφαλίσω ότι θα έχουμε μια έκθεση που μπορεί να αντανακλά νομίζω μια ευρύτατη πλειοψηφία από πλευρά του Ευρωκοινοβουλίου. Τουλάχιστον αυτό ελπίζω. Κάποια από τα κυριότερα σημεία που συζητήθηκαν. Προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε την ίδια κατεύθυνση που και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Δηλαδή, σε σχέση με τις συστάσει και τις συζητήσει για την έκθεση ετήσια προόδου και σε σχέση με το τι θα έπρεπε να, κάνει, να γίνει και από πλευρά Ευρωβουλή. Ξεκινάμε με κάποιες γενικές κοινέ παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να σημειώσουμε ότι σήμερα έχουμε μια πολύ ευάλωτη, ευαίσθητη κατάσταση έχουμε την απαρχή μιας οικονομικής ανάκαμψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά απομένουν πολλά προβλήματα όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, την υλοποίηση και εφαρμογή διαθωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, αλλά και το θέμα της υπερχρέωσης των κρατών μελών. Το χρέος εδώ είναι μια επιβάρυνση, ένα βάρος. Προγράμματα προσαρμογής που δίνουν καρπούς από τα κράτη-μέλη πρέπει πολύ προσεκτικά να εποπτεύονται και να λειτουργήσουν. Και εδώ και σε σχέση με την αλληλεγγύη και τους όρους και προϋποθέσεις που θα πρέπει να ισχύσουν, το, αναφέρ, το ανέφερε αυτό ο κύριος Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κύριος Ντράγκη, αλλά και την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης, όπου κάποια στοιχεία εξακολουθούν να απουσιάζουν και πρέπει να γίνει ταχαίως ε, να σημειωθεί πρόοδος επ' αυτών. Ως προς αυτά η έκθεση πραγματικά αντανακλά αυτά τα τρία ή τέσσερα κυριότερα στοιχεία για την υλοποίηση διαθωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Μακροπρόθεσμα η προσπάθεια επενδύσεων και διάθεσης κεφαλαίων για τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κίνητρα όσον αφορά φορολογικά συστήματα, ο προστατευτισμός από πλευρά των κρατών μελών μέσα από την παγκοσμιοποίηση φυσικά που βλέπουμε ότι αποτελεί μέρο τη λύσεω ε, για ε, τι οικονομίες μα ε, για τι αγορέ εργασία. Πρέπει να προαγάγουμε την κινητικότητα μεταξύ κρατών μελών για του εργαζόμενου, με την κινητικότητά του και όλα αυτά να οδηγήσουν σε μια κατάσταση όπου ευελπιστούμε ότι σταδιακά θα μπορέσουν να αρθούν τα προβλήματα μη ισόρροπων σχέσεων που εξακολουθούν εξακολουθούν να εφίστανται μεταξύ των οικονομιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα σήμερα. Κάνουμε και κάποιε παρατηρήσει για τη μείωση του χρέου, όχι μόνο στο δημόσιο χρέο, αλλά και στο ιδιωτικό χρέο. Και πρέπει τώρα να υπάρξει και οικονομική ανάκαμψη και ε, ανάπτυξη και συγκεκριμένα μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν. Και τέλο, εξίσου σημαντικό έχουμε και θέματα για την καταπολέμηση τη φοροδιαφυγή. και τέλο, εξίσου σημαντικό ενίσχυση, ενδυνάμωση της ε, ε, δημοκρατική λογοδότηση. Αυτό ήταν πάντα ένα κέριο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εντάσσεται και σε αυτή την έκθεση. Δεν υπησερχόμεθα σε συζήτηση και επίση συμφωνήθηκε μεταξύ των σχεδόν εισηγητών στι πρώτε συναντήσει να έχουμε ε, ε, εξειδικευμένα παρατήματα σε σχέση με τις λεπτομέρειες. Έχουμε έτσι συνοπτικά μια τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που νομίζω το μέγιστο αριθμό μελών μπορεί να συμπεριλαμβάνει και σε σχέση με θέματα που μπορεί να τεθούν ελπίζω ότι όλα αυτά θα μπορέσουν να ληφθούν υπόψη με παρατηρήσεις και σχόλιά σας για την τελική μορφή της έκθεσης που θα λάβει. Ευχαριστούμε κύριε Σίγητα. Και τώρα από πλευρά και όντω εισηγητού του ΕΛΚΑ, από πλευρά μου θα ήθελα πρώτα απ' όλα να τονίσω το μεγάλο έργο και θετικό έργο που επετέλεσε ο κύριος Ντεμπάκερ ε, εισηγητή σε αυτό το σχέδιο, για αυτό το σχέδιο έκθεσης κατάφερε να ισορροπήσει τα μελήματά μας και τα διαφορετικά θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν τους επόμενους μήνες. Και επιπλέον σε σχέση με αυτά τα οποία είπε ο κ. Ντεμπάκερ θα ήθελα να προσθέσω κάτι ή να τονίσω πρώτον τη σπουδαιότητα <clears throat> το ότι βλέπουμε να ε, φως στην άκρη του τούνελ επιτέλους αλλά ακόμα πολλά απομένουν και πρέπει να γίνουν και αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ακριβώς αυτή η πτυχή. Πολλά απομένουν και πρέπει να γίνουν. Υπάρχουν κάποια θετικά μηνύματα που μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε το 2014, το επόμενο έτος, με κάποια αισιοδοξία. Έχει τεράστια σημασία όμως να εξηγιανθεί η οικονομική κατάσταση και να παγιωθεί. Για να εξηγιανθεί και να παγιωθεί, εμπεδοθεί η οικονομική κατάσταση, έχει κέρια σημασία, πιστεύω, να τονίσουμε το ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και συγκεκριμένα, ως ε, ήθιστε να ε, λέμε, να διασφαλίσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ότι θα έχουν πρόσβαση σε πιστώσεις και δάνεια συγκρίσιμους όρους ε, στην ε, ζώνη ευρώ μεταξύ των διαφορετικών κρατών. Να μπορούν να χρηματοδοτηθούν δηλαδή ανάλογα με την οικονομική τους κατάσταση ε, και τις ανάγκες τους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι λόγω της έδρας τους μόνο. Και γι' αυτό είναι σημαντικό επίσης στην έκθεση να τονιστεί ή να ζητηθεί και να υλοποιηθούν τα μέτρα τα οποία έχουν προταθεί και βρίσκονται στο τραπέζι. Είναι σημαντικό να τονίσουμε και να ζητήσουμε ένα πιο δραστήριο ρόλο για επενδύσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σε όλα όσα αφορούν τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μπορεί να γίνει αυτό και υπήρξαν προτάσεις ε, ε, που τέθηκαν στο τραπέζι για να γίνουν περισσότερα και πιστεύουμε ότι περισσότερα μπορεί να πράξει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επίσης. Και μια άλλη πτυχή που θα ήθελα να υπογραμμίσω χωρίς αμφιβολία είναι η καταπολέμηση της ανεργίας. Η καταπολέμηση ιδιαίτερα της ανεργίας των νέων που πρέπει να είναι κύρια προτεραιότητα χωρίς καμιά αμφιβολία για όλους μας. Ως προς αυτή την πτυχή απευθύνεται έκκληση ώστε τα κονδύλια τα οποία αφορούν την εγγύηση, το εγγυητικό ταμείο, εγγυοδοτικό ταμείο για τους νέους να μπορούν να φτάσουν στους αποδέκτες και να λειτουργήσουν τα κράτη-μέλη με αυτά το δυνατόν ταχύτερα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την κατάσταση αυτή να παραμένουν οι νέοι επί μεγάλο χρονικό διάστημα ψάχνοντας για δουλειά και όντας άνεργοι. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε και να ληφθούν υπόψη τα προβλήματά τους και να αναζητηθούν, πρέπει να αρχίσουμε να αναζητούμε λύσεις στα προβλήματά τους με το πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ένας από τους πιο σημαντικούς πυλώνες, όχι ο, η μόνη, ο μόνος άξονας, αλλά ένας από τους κύριους άξονες είναι το Ταμείο Εγγύησης για τους Νέους και να μπορέσουμε να δράσουμε με αυτό αποτελεσματικά. Και μέσα στο πλαίσιο της ε, χρηστής διακυβέρνησης τονίζω τη σπουδαιότητα του μέσου ανταγωνιστικότητας ε, ε, με τα αγγλικά αρχικά του στο ακρόνιμο και έτσι με αυτό θα πρέπει να πετύχουμε τη σύγκληση των οικονομικών επιδόσεων και των εισοδημάτων των κρατών μελών ώστε να επανορθώσουμε, να διορθώσουμε τις μη σχέσεις και δομικά που υπάρχουν σε σχέση με αυτά τα θέματα. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία στοιχεία που ως και ό,τι θα ήθελα να αναφέρω. Και δίνω αμέσως τώρα τον λόγο στη συνέχεια στον κύριο Ονιόκ που αντικαθιστά την κυρία Σκιώδη εισηγήτρια των σοσιαλιστών σε αυτό το θέμα. Κυρία Ποδήματα, παρακαλώ. Σε ευχαριστώ, Πάμπλο. Θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ σε αυτά τα οποία θα έλεγε η Ιάννη, η συνάδελφός μου. Θα σας διαβάσω βασικά το σημείωμα το οποίο μου έδωσε η κυρία Ποδηματά αναφέρει ότι ε, είναι δυνατόν να συζητηθούν διάφορα σημεία της έκθεσης αυτής. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία θα ψηφιστεί, θα πρέπει να δώσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είμαστε ικανοποιημένοι όσον αφορά τη δημοκρατική νομιμότητα και όσον αφορά επίσης κατευθυντήρες γραμμές. Μολονότι ο εισηγητής έκανε σημαντικές προσπάθειες και στέλνει κάποια θετικά μηνύματα, παρόλα αυτά η έκθεση δεν αντικατοπτρίζει την επιθυμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη κοινοτική μέθοδο, αλλά και μια πραγματική δημοσιονομική εξυγίανση η οποία ευνοεί την ανάπτυξη. Τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής θα πρέπει να εναρμονιστούν με τους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα πρέπει να αναβαθμιστεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα προγράμματα μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να βασίζονται στις κατευθύνσεις γραμμές σύγκλησης. Η κυρία Ποδηματά επίσης δεν εμπιστεύεται ιδιαίτερα το όλο σύστημα σύμπραξης συμβάσεων, δεν χρειαζόμαστε ένα σύστημα ex post για την αξιολόγηση των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή τη στιγμή συμμετέχει στην Τρόικα. Πράγμα το οποίο το βλέπουμε και στην έκθεση Φερέιρα, η οποία έχει ήδη εγκριθεί. Όσον αφορά την οικονομική πολιτική, χρειαζόμαστε μια δημοσιονομική εξυγένση η οποία ευνοεί την οικονομική ανάπτυξη. Αυτό παραμένει απλώς ευσεβής πόθος αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει επίσης να ακολουθούμε περισσότερο τις προτεραιότητες στρατηγικής Ευρώπη 2020. Δεν θα πρέπει να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά όσον αφορά τις διάφορες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, σοβαρά οικονομικά προβλήματα θα πρέπει τα προγράμματα προσαρμογής να γίνονται αποδεκτά και από, τον, από το κοινό, από τον πληθυσμό της κάθε χώρας, να εμπνέονται από την κοινωνική δικαιοσύνη. Θα πρέπει να υπάρχει ένας ισότιμος επιμερισμός όλων των προσπαθειών που γίνονται από τους Ευρωπαίους πολίτες και ότι ο σύστατο μέσο θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη φορολογία και μόνο ο σύστατο μέσο. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις στην έκθεση Κλέβα θα πρέπει επίσης να έχουμε συγκεκριμένους δείκτες καταμέτρησης της πρόοδου των κρατών μελών και ότι θα πρέπει πάλι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο να ακολουθεί περισσότερο τους στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020. Θα πρέπει επίσης να έχουμε συγκεκριμένους στόχους για την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων. Η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης. Παραλείπω το σημείο αυτό γιατί δεν είναι ο Λεωμιλητής... η δημοσιονομική εξυγίανση θα πρέπει να επιτρέπει και τις επενδύσεις στο δημόσιο τομέα. Χρειαζόμαστε ένα νέο πράσινο New Deal για να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές και κάτι που θα μπορούσε να δημιουργήσει και οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε επίσης την φτώχεια, την ένδια και την ανισότητα και δεν θα πρέπει επίση να μειώνονται περαιτέρω οι μισθοί, να υπάρχει επίση ελάχιστο μισθό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά λέει στο σημείωμά τη κυρία Άννη Ποδηματά. Green... Εξ ονόματο των Πρασίνων, ποιο είναι εδώ, δεν βλέπω κανέναν, λέει ο Πρόεδρο. Συνεχίζουμε. Εξ ονόματο του ECR, ο σκιώδη συζητητή είναι ο κύριο Έπινγκ, αλλά εσεί, κύριε Στρέτσικ θα τον αντικαταστήσετε, έτσι δεν είναι, έχετε το λόγο. Ακριβώς κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Σέπινγκ χρειάστηκε να παραμείνει στι Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως, μου ζήτησε να σας διαβάσω τις παρατηρήσεις του. Έχω εδώ ένα ολόκληρο κατάλογο, 8-9 παρατηρήσεις έχει να κάνει ο κύριος Σέπινγκ. Θα μπορούσαμε να τις χωρίσουμε σε δύο τμήματα. Στο πρώτο τμήμα ο κύριος Σέπινγκ συμφωνεί με τον κύριο Μπάκερ, με την έκθεσή του δηλαδή. Καλύτερα να σα διαβάσω τα όσα γράφει ο κύριο Σέπινγκ στο σημείωμά του. Πρώτον, θέλει να ευχαριστήσει τον εισηγητή για την επικοδομητική προσέγγιση στην έκθεσή του, καθότι προσπάθησε να βρει κάποια κοινά επιχειρήματα και δεν επέμεινε στα σημεία αυτά τα οποία μας διαχωρίζουν. Είμαστε ικανοποιημένοι με το σχέδιο έκθεσης του κυρίου Ντεμπάκερ, γιατί αναγνωρίζει το ότι η κρίση δεν έχει ακόμα παρέλθει και ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε τη δημοσιονομική εξυγίανση η οποία θα ευνοεί την οικονομική ανάπτυξη και να συνεχιστούν βέβαια και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Υποστηρίζουμε εμεί τι επενδύσει πρέπει να γίνουν στον τομέα τη έρευνα και τη ανάπτυξη και τη εκπαίδευση. Θεωρούμε ότι ο ξεχρονισμό ε, των συστημάτων κοινωνική ε, υποστήριξη και υγειονομική περίθαλψης είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να έχουμε έναν πιο αποτελεσματικό δημόσιο τομέα. Επίσης υποστηρίζουμε τα όσα λέγονται για την μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδίως για την πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πραγματικά θέλουμε να ανακάμψει η πραγματική οικονομία και θέλουμε να δημιουργήσουμε μια, βασι... μια σταθερή, ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι τα σημεία με τα οποία συμφωνούμε με το σχέδιο έκθεση του κ. Ντεμπάκερ. Περνάμε τώρα στο άλλο τμήμα. Δεν συμφωνούμε με το ότι τα προγραμματα υποστήριξης υποστήριξη ορισμένα κράτη-μέλη θα πρέπει να υπέλθουν στο κοινοτικό πλαίσιο. Επίσης ε, δεν πιστεύουμε ότι η ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης ε, είναι αυτό το οποίο θα πρέπει πραγματικά να προωθήσουμε όταν υφίστανται τόσα πολλά εκκρεμή ακόμα ζητήματα τα οποία πρέπει κατά προτεραιότητα να επιληθούν προτού περάσουμε σε μια βαθύτερη ένωση. Ο κύριος Σέπινγκ επίσης τονίζει ότι το ευρωπαϊκό εξάμεινο που γίνεται κάθε χρόνο και ξεκινάμε την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης είναι ένα τεχνικό μέσο δημοσιονομικού συντονισμού και όχι μία, ένας κατάλογος κάποιων πολιτικών στόχων. Νομίζω, νομίζω τουλάχιστον ο κύριο Σέπινγκ ότι ο, οποιοδήποτε αναφορές γίνονται στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση πρέπει να γίνει σε κάποια άλλη έκθεση και όχι σε αυτήν εδώ. Ευχαριστούμε. Εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ενωτικής Αριστερά δεν βλέπω κανέναν. Συνεπώς, αρχίζει η συζήτηση με τους υπόλοιπους. Η κυρία Λούλινγκ. Παρακαλώ, κυρία Λούλινγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Διάβασα το σχέδιο αυτό πρότασης ψηφίσματος. Γενικά μιλώντας, είναι καλό η διατύπωση όμως είναι αρκετά ασαφής. Σε διάφορα σημεία μάλιστα δεν κατάλαβα. Γι' αυτό έχω ερωτήσεις. Σημείο 2. Εδώ ζητάμε μείωση των τιμών και προσαρμογή στην παραγωγικότητα του εργατικού κόστος. Δηλαδή να προσαρμόσουμε το εργατικό κόστος στα επίπεδα που συμβαδίζουν με την παραγωγικότητα, αυτό τι σημαίνει. Δεν ξέρω αν υπάρχει βέβαια ακόμα στο Βέλγιο αυτόματη αναπροσαρμογή στο δίχτυ τιμών, όποια και αν είναι τα αποτελέσματα στην παραγωγικότητα. Επίσης, λέτε ότι πρέπει να γίνουν πιο ανταγωνιστικές οικονομίες, ε, ανάπτυξη, εννοείται κανένας δεν είναι κατά. Κανείς δεν είναι κατά του πέντε Φυσικά και πρέπει να μειωθεί το χρέος. Στο σημείο 7 όμως, λέτε, συγχαίρει τις αρχές των κρατών μελών που εφάρμοσαν επιτυχώς προγράμματα προσαρμογής. Ποιες χώρες μέλη συγχαίρεται δηλαδή για να καταλάβω. Πολύ θα ήθελα να το ξέρω. Γιατί εγώ έρχομαι από μια χώρα όπου επαναλαμβάνουμε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου τις ίδιες συστάσεις εδώ και χρόνια. Ότι δεν ε, ακολουθήσαμε τις συστάσεις και τα λοιπά, αλλά μετά δεν γίνεται τίποτα. Το Συμβούλιο τελικά επικυρώνει τις συστάσεις και οι κυβερνήσεις κάνουν ό,τι θέλουν. Αδιαφορούν. Εμείς υπενθυμίζουμε γίνονται ίδιες συστάσεις συνεχώς. Επίσης στο σημείο 11 λέτε ότι πρέπει να μειωθούν οι φόροι και οι σφορέ οι ασφαλιστικέ. Μα ξέρετε ότι έχουμε προβλήματα χρηματοδότησης ορισμένων ασφαλιστικών ε, ταμείων. Πώς μπορούμε να μειώσουμε τις εισφορές της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μου, για παράδειγμα. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν καταλαβαίνω πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να αυξηθούν για να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση των συντάξεων. Λέτε επίσης στο σημείο 13 και εδώ συμφωνώ απόλυτα πολύ σωστά τα λέτε στο σημείο 15 όμως μιλάτε και πάλι για την φορολογία που αποτελεί μια επιβάρυνση. Εσείς εδώ θέλετε δηλαδή αύξηση του ΦΠΑ. Στο σημείο 19 επίσης λέτε ότι πρέπει να υπάρξει μια κοινή αγορά εργασίας και μια πολιτική σύγχρονης μετανάστευσης. Αυτό το σύγχρονη δεν μου αρέσει. Ο καθένας το ερμηνεύει διαφορετικά. Τι εννοείτε εσείς με τη σύγχρονη πολιτική μετανάστευση, με τι κριτήριο δηλαδή. Σημείο 28. Εδώ εκφράζεται την ανησυχία, διότι μόνο δύο κράτη-μέλη πέτυχαν το μεσοπρόθεσμο στόχο. Ποιες είναι αυτές οι δύο, θέλω να ξέρω. Τέλος, για το σημείο 29. Εδώ λέτε ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο δεν πρέπει κατ' ουδένα τρόπο να θέσει κίνδυνο τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων και υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να υπάρξει σαφής διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών μελών. Αν όμως λέτε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και για χρόνια μια χώρα δεν συμμορφώνεται στις συστάσεις, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, τότε οι χώρες μέλη με αυτή τη διατύπωση τι καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνουν ότι μπορούν να συνεχίσουν να μην συμμορφώνονται. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Στη χώρα μου αυτό γίνεται. Το κοινοβούλιο όταν αναλύει τις συστάσεις ακόμα και στις ειδικές επιτροπές, έρχονται υπουργοί και λένε ότι οι συστάσεις δεν ισχύουν. Το Κοινοβούλιο λέμε εδώ δεν υπάρχει τίποτα καινούριο, γίνεται η ίδια σύσταση που είχαμε και πέρυσι και πρόπερσι. Όταν για τρία χρόνια η σύσταση είναι ίδια, σημαίνει ότι δεν έκαναν τίποτα, ότι δεν διόρθωσαν, δεν συμμορφώθηκαν με τις συστάσεις. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να είμαστε πιο συγκεκριμένοι εδώ και να μην έχουμε τέτοιες διατυπώσεις που αφήνουμε τις χώρες μέλη να νομίζουν ότι μπορούν να διαφορίζουν πλήρως για τις συστάσεις όσον αφορά το ευρωπαϊκό εξάμενο, ότι τις γράφουν στα παλιά του τα παπούτσια δηλαδή, για συγγνώμη για την έκφραση. Ευχαριστούμε κυρία Λούλινγκ. Η κυρία Μπερές που είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης. Παρακαλώ κυρία Μπερές. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εδώ δεν παίρνω το λόγο ως πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης, παρόλο που στην Επιτροπή αυτή όπου συμμετέχει και ο εισηγητής της Οικονομικής Επιτροπής ε, δείχνει ότι υπάρχει μια σχέση. Για την έκθεση τώρα του συναδέλφου Ντεμπάκερ. Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια για την παράγραφο αριθμός 30 Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε για τα Εθνικά Κοινοβούλια να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη. Αλλά εδώ, αν θέλουμε να περάσει το μήνυμα αυτό, πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο σκέψης του Συμβουλίου για τον ενιαίο μηχανισμό εξυγένσης, που κινδυνεύει να ενισχύσει το έλλειμμα αυτό. Συνεπώς, για να περάσει αυτό το μήνυμα πρέπει να το συμπληρώσουμε βάσει της πρόσφατης επικαιρότητα, δηλαδή των εργασιών του ΕΚΟΦΗΜ. Απ' την άλλη όμως, για την παράγραφο 21 που αναφέρεται στην αξιολόγηση, νομίζω ότι εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Λέτε ότι η εξέταση δεν είναι αρκετά λεπτομερής, αλλά δεν αναφέρεστε στο περιεχόμενο. Τι μέσα λοιπόν έχει το Κοινοβούλιο για να επηρεάσει. Βλέπουμε, το βλέπουμε εδώ, πόσο λίγοι είμαστε, ελάχιστα ενδιαφέρονται. Άχιστοι θα ασχοληθούν με τη συνέχεια. Κάποιοι θέλουν έναν κώδικα σύγκλησης. Δεν ξέρω, δεν είναι δυνατόν να κερδίσουμε καμία μάχη αν αλλάζουμε θέση κάθε τρεις και λίγο. Το Κοινοβούλιο λέει ότι στο σημερινό στάδιο, έτσι όπως έχει διακυβέρνηση στην Ευρωζώνη και την ΟΝΕ, έτσι ως έχει σήμερα, το θέμα της ετήσιας εξέτασης της ανάπτυξης είναι σημαντικό για να οργανωθεί η δημοκρατική συζήτηση και ότι το μέσο που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δράσει σαν να είναι περίπου συνομοθέτης επ' αυτού, κάτι με το οποίο είχαμε συμφωνήσει εδώ και καιρό στην αρχή της θητείας, ε, λοιπόν, τότε πρέπει την ετήσια εξέταση της οικονομικής ανάπτυξης πρέπει να την εξετάσουμε σαν να πρόκειται για νομοθετικό κείμενο και εμείς οι ίδιοι να μπαίνουμε στη λεπτομέρεια όσον αφορά τις συστάσεις προς τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό και βλέπω εδώ αντίφαση και λυπάμαι ότι εξήγηση και αν δώσετε λυπάμαι που δεν υπάρχει παράρτημα που να επιτρέπει με σαφήνεια να προωθηθεί η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η συμμετοχή του στην εξέταση της ετήσιας οικονομικής ανάπτυξης. Δεύτερον, η ισορροπία του κειμένου ανάμεσα στην διαρθρωτική μεταρρύθμιση και την ανάγκη για εξοικονόμηση πόρων. Μπορεί να το διάβασα βιαστικά, αλλά με εκπλήσει γιατί βλέπω ότι η έλλειψη δημοσίων ε, και ιδιωτικών επενδύσεων που δεν ε, εντοπίζονται στην ετήσια εξέταση της οικονομικής ανάπτυξης δεν εντοπίζονται ούτε εδώ με σαφήνεια. Το Γερμανικό Ινστιτούτο, δηλαδή όσον αφορά τις δημόσιες επενδύσεις στη Γερμανία, αναφέρεται σε αυτό. Ξέρουμε ότι και στη Γαλλία δεν υπάρχουν αρκετέ επενδύσεις. Άρα λοιπόν πέρα από τις διορθωτικές μεταρρυθμίσεις υπάρχει και αυτό. Και οι διορθωτικές μεταρρυθμίσεις δεν νομίζω ότι φτάνουν για να επιστρέψουν οι επενδύσεις. Χρειαζόμαστε και το ένα και το άλλο. Πρέπει να εντοπιστεί η έλλειψη των επενδύσεων αυτών και μετά να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί. Τέλος, όσον αφορά την φορολογία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μερικές φορές είναι πολύ διστακτική σε συστάσεις στον τομέα αυτό. Παρόλο που μερικές χώρες ανάμεσα στην φορολογία κεφαλαίου, εργασίας και οικολογική θα έπρεπε να εξεταστούν πιο συγκεκριμένα. Διαφωνώ με την κυρία Λούλινγκ ελαφρώς η φορολογία εργασίας και ΦΠΑ μπορεί να μην είναι κάτι επιθυμητό, η φορολογία της εργασίας όμως είναι κάτι το οποίο έτσι καλώ πρέπει να τεθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε όμως να το κάνουμε μεταφέροντας την προς την κατανάλωση, γιατί μία από τις λειτουργίες της φορολογίας αυτής της εργασίας είναι ακριβώς το ότι δεν έχει επιτευχθεί. Έπειτα, οικολογική διάσταση. Για να λυθούν υπόψη οι πιο εύθραυστες κοινωνικά καταστάσεις, είναι και αυτό κάτι που πρέπει να, πάνω στο οποίο πρέπει να επεκταθούμε περισσότερο. Έπειτα η φόρο διαφυγή είναι και αυτό ένα θέμα που πρέπει να αναφέρουμε. Επιμένουν λοιπόν για τα θέματα των επενδύσεων πρώτα απ' όλα και των παραρτημάτων. Έπειτα διατησία ανάμεσα στην ε, φορολογική μεταρρύθμιση και τις επενδύσεις. Εδώ διαπιστώνουμε να δείτε μια συζήτηση η οποία έχει αρχίσει εδώ και δύο χρόνια. Οι επιπτώσεις δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Είναι η συζήτηση που κάνει και το Διεθνές Μεσοκό Ταμείο για τους πολλαπλασιαστές, τους δείκτες δηλαδή σε σχέση με την οικονομική λιτότητα καθημερινά βλέπουμε με στοιχεία από τους εμπειρογνώμονες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως δεν θέλει να πάρει μαθήματα από αυτά. Ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θελήσει. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Μπερές. Σας ευχαριστούμε πολύ επίσης που διευκρινίσατε για το ότι δεν μιλάτε ως πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης. Ο κύριος Δεμπάκερ έχει το λόγο. Σας Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τα μέλη για τα σχόλια που έκαναν. Για τα σχόλια στην έκθεση. Και για να είμαι σύντομος και αναφερόμενο σε κάποια από τα σημεία που εξετέθησαν. Και για την κυρία Ποδήματα αυτά που ακούστηκαν και πράγματι για την ε, δημοκρατική νομιμότητα. Εδώ πρέπει κάποια πράγματα να αποσαφινιστούν στο πλαίσιο της έκθεσης. Και είμαι πρόθυμος να δω πώς μπορεί να γίνει αυτό και στις διατυπώσεις που θα επιλεγούν Πιστεύω ότι πραγματικά αυτό πρέπει και μπορεί να είναι ένα από τα ισχυρά σημεία αυτής της έκθεσης και πρέπει να συνεχίσουμε το έργο μας, την εργασία μας προς αυτή την κατεύθυνση αποσαφήνισης και εξετέθησαν και οι τοποθετήσεις των διαφορετικών ομάδων. Είχαμε αυτή τη συζήτηση δύο-τρεις φορές ε, και καταλήγουμε στα ίδια σημεία κάθε φορά. Το πρόγραμμα το οποίο ακολουθήθηκε από πλευρά ε, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ασκώντας και μεγαλύτερη πίεση στα κράτη-μέλη ώστε να διασφαλιστεί ότι πραγματικά θα υπάρξει η αηφορία και ταυτόχρονα θα επιτευχθεί η ε, υλοποίηση διαθωτικών ε, ε, μεταρρυθμίσεων στα κοινωνικά συστήματα για την καινοτομία. Όλα αυτά είναι θετικά ή όχι. Είναι και κάπως ιδεολογική η συζήτηση και ίσως και ιδεολειπτική και προσπαθεί η έκθεση να γεφυρώσει τις διαφορετικές απόψεις δεν έχει καταδειχθεί επαρκής ε, αξιοπιστία σε σχέση με τις συστάσεις που έχουν διατυπωθεί. Και είναι και κάποια από τα θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της έκθεσης. Αν θέλουμε να στεφθεί με επιτυχία το ευρωπαϊκό εξάμεινο και να αυξηθεί η εμπιστοσύνη, ευρωπαϊκή εμπιστοσύνη, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να δράσουν και από πλευρά τους. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει συμφωνία επί κάποιων συστάσεων και μετά <clears throat> να λέγεται ότι αυτά πρέπει να γίνουν από πλευρά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή από ε, πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε συμφωνήσει, ε, υπάρχει συμφωνία για το six και τι διάφορε άλλε προτάσει. Δώσατε την έγκρισή σα ε, σε αυτή την ε, ετήσια έκθεση. Έτσι λοιπόν και από πλευρά των κρατών μελών η εμπλοκή θα έχει μεγάλη σημασία. Και εδώ αντανακλώνται και τα σχόλια της κυρίας Λούλινγκ επ' αυτού και εντάσσονται σε ένα σφαιρικότερο πλαίσιο. Δεν θα επισέθω σε λεπτομέρειες όπως για παράδειγμα για το άρθρο 2. Είπαμε σε σχέση με αυτό ότι πρέπει να προαχθεί περαιτέρω η ανταγωνιστικότητα και το ουσιαστικότερο μήνυμα σε αυτό είναι ότι αν το μισθολογικό κόστος αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό από την παραγωγικότητα, τότε χάνουμε ανταγωνιστικότητα. Όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα, χάνουμε έδαφος. Είναι ένας βασικός ε, νόμος. Πρέπει αυτά να μπορέσουν να βαίνουν εκ για να υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη. Και για το άρθρο 7 υπάρχουν κάποιες ε, χώρες που μπόρεσαν να επιστρέψουν στις αγορές όπως η Ιρλανδία για παράδειγμα υπάρχει αυτή η αναφορά και υπάρχει και η διευκρίνηση για το, ε, ε, το τι συνέβη και τι ε, ακολουθεί και νομίζω υπάρχει μια γενικότερη τοποθέτηση γιατί δεν ξέρουμε αν κάποια χώρα μπορεί και εκείνη μελλοντικά να εξέλθει από το πρόγραμμα και για το άρθρο 28 υπάρχουν φυσικά χώρες που από την άλλη πλευρά έχουν και καλές επιδόσεις και βρίσκονται στα όρια τα οποία έχουν επιβληθεί μέσω του Six Pack ή του Συμφώνου Σταθερότητας. Η Εστονία και η Γερμανία είναι σε αυτή την κατηγορία. Υλοποιούν τις υποχρεώσεις ε, που ε, είχαν διαπιστωθεί και είχαν καθοριστεί και έτσι λοιπόν σε σχέση με το να ονοματίσουμε συγκεκριμένες χώρες αναφέρουμε αυτές τις δύο εδώ σε αυτό το σημείο και για την απλούστευση, απλούστευση των φορολογικών συστημάτων και την ε, μετάθεση ε, κέντρου βάρους. Ε, βλέποντας τα υπό ένα ευρύτερο πλαίσιο θα πρέπει η φορολόγηση να απόσχει, να αποστασιοποιηθεί από το μισθολογικό κόστος. Δεν είναι το μόνο στοιχείο το μισθολογικό κόστος. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη και τα θέματα και τα περαιτέρω θέματα. Πρέπει να μεταβούμε από την φορολόγηση της εργασίας και σε φορολόγηση άλλων παραμέτρων ώστε με διάφορα κριτήρια να μπορούν μέσα σε ένα σφαιρικό σύστημα να λειτουργήσουν αυτές οι αρχές καλύτερα και το ανέφερε και η κυρία Λούλινγκ. Φυσικά με ένα γυράσκοντα πληθυσμό θα πρέπει να γίνει συζήτηση για τα θέματα κοινωνικής ασφάλισης και να δούμε πώς θα χρηματοδοτηθούν μελλοντικά. Αλλά είναι σημαντικό να έχουμε μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα που θα πετύχουμε και περισσότερο μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που θα ε, συμμετέχουν στην αγορά εργασίας ε, στο ασφαλιστικό σύστημα και να δούμε πώς θα μπορέσουν τα συστήματα φορολόγησης να είναι λειτουργικά. Και ίσως κάποιες παρατηρήσεις τώρα και για τα άλλα θέματα τα οποία αναφέρθηκαν από την κυρία Μπερές ο λόγος για τον οποίο δεν κάναμε το παράρτημα είναι διτός. Αφενός δεν υπάρχει πολιτική πλειοψηφία που να εγκρίνει αυτό από πλευράς αυτού του Κοινοβουλίου και το είδαμε και στη συζήτηση για το εξάμεινο και δεύτερον πιστεύω ότι αν θέλουμε να το κάνουμε αυτό πρέπει να το κάνουμε σοβαρά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να έχει στη διάθεσή της πολλές αναλύσεις ε, για τα όσα τεκταίνουν στα κράτη-μέλη και αν θέλουμε να επαναλάβουμε αυτό το εγχείρημα εμείς πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτό το εγχείρημα με σοβαρότατο τρόπο δεν θα, θε, δεν θα επιτρέψω με κανένα τρόπο να υπάρξουν παρατήματα όπου ευχολόγια και πολιτικές επιθυμίες των κρατών μελών ε, θα εντάσσονται σε αυτά τα παρατήματα. Δεν είναι καθόλου αναγκαίο, είναι απόλυτα περιττό αυτό. Και δεν υπάρχει και πολιτική πλειοψηφία που να εγκρίνει από το Κοινοβούλιο να γίνει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ρωτώ, ρώτησα τους ευ, ε, αν θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και να εγκρίνουμε το παράτημα. Και η συντριπτική πλειοψηφία ακόμα και των πρασίνων ήταν να μην υπάρξει ένα τέτοιο παράτημα παράρτημα. Σέβομαι την βούληση λοιπόν της πλειοψηφίας και κατανοώ ότι είναι κάπως απογοητευτικό ίσως για την ομάδα σας και σε σχέση με τις λεπτομέρειες και για τα θέματα επί των οποίων εργαζόμαστε για αυτή την έκθεση με τους κοιόδης εισηγητές είναι πραγματικά νομίζω σε πολύ διάφανο τρόπο για, ε, που καθορίζουμε αυτά τα στοιχεία. Η άλλη συζήτηση και πάλι όπως προανέφερα στην αρχή είναι τα θέματα οικονομικής ε, ε, προσέγγισης από πλευράς ιδεολογίας δείκτες για την εξαίρεση για παράδειγμα όσον αφορά αφορά την ε, λιτότητα. Αναφέρονται κάποια θέματα σύντομα στην έκθεση, αλλά δεν είναι αυτή η ουσία τη συζήτηση. Στην ουσία της όλοι συμφωνούμε επ' αυτού είναι πώ μπορούν τα κράτη-μέλη να οδηγηθούν στην ανταγωνιστικότητα, να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία, να δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση και εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να δώσουμε κίνητρα στι μικρομεσαίες επιχειρήσει ώστε να σημειωθεί ανάπτυξη και ε, να υπάρξει ανάπτυξη τη οικονομία. Όλα αυτά τα θέματα εξετάζονται στην έκθεση και προσβλέπω στο να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση με όλους σας στο μέλλον και να καταλήξουμε σε μια με μεγάλη πλειοψηφία που θα εγκριθεί έκθεση και υπάρχουν θέματα που είναι πολλά, πολύ περισσότερο ε, ανεπτυγμένα από, ε, από την Επιτροπή Οικονομικών Νομισματικών Θεμάτων ώστε να μπορέσουν ε, οι δύο εκθέσεις να βαίνουν εκ παραλίλου. Θα ήταν κακό μήνυμα να έχουμε δύο εκθέσεις οι οποίες αποστασιοποιούνται μεταξύ τους και βαίνουν προς διαφορετική κατεύθυνση. Θα πρέπει να βαίνουν εκ παραλίλου. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντεμπάκερ. Η 9 Ιανουαρίου είναι η ημερομηνία καταβολής των τροπολογιών. Θα ψηφίσουμε στις 13 Ιανουαρίου στην Επιτροπή μας, αφού εξετάσουμε τις τροπολογίες, και στην Ολομέλεια θα ψηφίσουμε το Φεβρουάριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώνται στο σημείο αυτό η συζήτηση. Αύριο το πρωί θα συνεχίσουμε με τον οικονομικό διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό Οικονομικών της Λιθουανίας. Η συζήτηση αυτή θα λάβει χώρα σε 9 ώρα το πρωί. Στην ίδια την αίθουσα. Πολύ ωραία λοιπόν, λίγη τη συνειδρίαση.